Good morning. Buenos Καλημέρα σας. Good morning. If you're Έχετε την καλοσύνη να καθίσετε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Με το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης σήμερα έχουμε μια πολύ ε, δραστήρια συνεδρίαση σήμερα μέχρι τις 12.30 και από τα 9.45 και πέρα έχουμε μια κρόση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και έχουμε και ψηφοφορίες 3 ε, με 4 και 4. Όσα μέλη λοιπόν ε, είχαν την καλοσύνη να έρθουν για το πρώτο θέμα της ημερήσια διάταξη σήμερα. Ας υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί και προχωρώ στο 11 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Δραστηριότητες της EASO. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα μας παρουσιάσει θα μας ενημερώσει για την ετήσια έκθεση ο κύριος Ρόμπερτ Βίσερ. Αυτή η έκθεση είναι η τρίτη και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της EACO στις 18 18-19 Ιουνίου φέτος και η ετήσια έκθεση αυτή Ε, παρουσιάζει τη γενική στρατηγική, ε, την, ε, την προγραμματισμό του προϋπολογισμού, τις διαστηριότητε της ΙΑΣΟ και ας ακούσουμε λοιπόν την εκτίση αυτή έκθεση, την εισήγησή του και μετά θα έχουμε το διάστημα των ερωταπαντήσεων. Ο κύριος Βίσερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκουμε ενώπιόν σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Στην ημερήσια διάταξη, όπως ανέφερε μόλις ο Πρόεδρος, βρίσκεται η ετήσια έκθεση της ΙΑΣΟ 2011. Ήταν ε, η πρώτη και όχι ολοκληρωμένη, διότι εγώ διορίστηκα 1η Φεβρουαρίου του 2011. Οπότε αυτή η έκθεση αντανακλά τους μήνες της θητείας, της θητείας μου. Επίσης, ε, όπως ζήτησε η Επιτροπή σας, θα αναφερθώ και στις δραστηριότητες του 2012 και στο πρόγραμμα εργασίας του 2013. Είναι ε, έγγραφα και προγράμματα ενημέρωση δηλαδή που μόλις εστάλει στην Επιτροπή σας ε, από τις υπηρεσίες μου. Όπως σας είπα αυτή τη στιγμή λειτουργούμε εδώ και 1,5 χρόνο, αρχίσαμε πέρσι και θα σας παρουσιάσω εν συντομία ε, τις δραστηριότητε και τα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα. Έχουμε τρεις γραμμές στήριξης μόνιμη στήριξη, ε, στήριξη σε κατάσταση έκτακτης ε, ανάγκης ε, και προσωρινή στήριξη, περιστασιακή στήριξη η πρώτη αντιπροσωπεύει τις κανονικές μας εργασίες, η δεύτερη μια κάπως προειδοποιητική ε, εργασία και, η τρίτη τις δραστηριότητε μας τις εξωτερικές. Ε, εργαζόμαστε όλοι στον τομέα του ασύλου και στη σύγκληση του ασύλου και της ε, μετανάστευσης και αυτή είναι μία θεμελιώδης ε, πτυχή των δραστηριοτήτων όλων των κρατών μελών. Γι' αυτό ε, στοχεύουμε στη διοργάνωση ε, εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στην εδραίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων έτσι ώστε σε όλη την επικράτεια της Ένωσης το, η κατάρτιση αυτή είναι ομοιόμορφη και ισοδύναμης για όλους. Ε, μπορέσαμε να οργανώσουμε πολλές συνεδριάσεις, ένα μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, μάλλον εκπαιδευτικών ε, ε, σεμιναρίων, 14 με 16 τέτοια εκπαιδευτικά σεμινάρια ή δραστηριότητες κατάρτισης θα διοργανώσουμε του χρόνου, έτσι το έχουμε προγραμματίσει και περιλαμβάνουμε και την Ελλάδα. Βεβαίως, μερικά από αυτά θα γίνουν στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάζουμε, εκπονούμε την βασική τεκμηρίωση την οποία χρειάζομαι, χρειαζόμαστε για να υποστηρίξουμε αυτά τα, αυτή την εκπαίδευση και η φιλοδοξία της υπηρεσίας είναι να καταλήξουμε σε μια κοινή έκθεση ασύλου μετανάστευσης από τις βασικές χώρες προέλευσης. Η πρώτη μας έκθεση για το Αφγανιστάν Δημοσιεύθηκε φέτος, η επόμενη θα δημοσιευτεί την, τον ερχόμενο μήνα και προγραμματίζουμε και πολλές άλλες εξέσεις να δημοσιευθούν, να συνταχθούν ε, μάλλον στο μέλλον. Αυτή είναι η βασική μας δραστηριότητα, η μόνιμη. Εν συνεχεία έχουμε την, ε, την στήριξη εκ, έκτακτης ανάγκης. Παραδείγματο χάρη είμαστε ήδη δραστηριοποιούμεσα στην Ελλάδα από το πρώτο εξάμεινο ε, του 2011 και μπορέσαμε από την πρώτη μέρα να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρμόδιες αρχές για την δημιουργία της υποδομής των υπηρεσιών που προβλέπει ο νόμος, που προβλέπουν οι νόμοι. Ε, έχουν δραστηριοποιηθεί ομάδες για το άσυλο, έχουμε αποστείλει εμπειρογνώμονες δικούς μας και έχουμε εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό των νέων υπηρεσιών και όταν έχουν διοριστεί περισσότερα στελέχη θα έχουμε τα προγράμματα έτοιμα, είναι ήδη έτοιμα τα νέα προγράμματα και ε, έχουμε ήδη εκδώσει εγχειρίδια εκπαιδευτικά και όλες τις πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης, τα COI. COI. Και επίσης ε, όλες αυτές τις, ε, την υποδομή που χρειάζεται για την εδραίωση και στελέχωση των κέντρων υποδοχής. Α. Επίσης, ε, ε, μπορούμε να υποστηρίξουμε χώρες ε, οι οποίες ε, δεν είναι χώρες μόνιμης στελέχωσης, οι χώρες που δεν εμπίπτουν στο μόνιμο πρόγραμμά μας, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Διότι αλλάζουν οι συνεργάτες μας και οι εταίροι μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία, οι βασικοί πυλώνες ε, της υποστήριξης της ΕΑΣΟ. Μόνιμη υποστήριξη, έκτακτη και ειδική περιστασιακή. Εκτός από αυτά, έχουμε αρχίσει και ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί, αν θέλει κανείς να προλάβει και να διορθώσει και να ε, υποστηρίξει ε, τα κράτη-μέλη με τρόπο χρήσιμο και ωφέλιμο, θα πρέπει αυτό να γίνεται νωρίς και όσο γίνεται ταχύτερα. Αυτό το σύστημα καταρτίζεται αυτό τον καιρό και ευτυχώς συμπίπτει και με τη συζήτηση που γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο για το άρθρο 31 του κανονισμού του Δουβλίνου. Συνδυάζουμε λοιπόν αυτές τις δύο δράσεις. Κατανοώ πλήρω και συνειδητοποιώ ότι το άρθρο 31 και ο κανονισμός του Δουβλίνου ακόμα δεν ισχύουν ε, θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης έχοντας υπόψη ότι μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά. Η έγκαιρη προειδοποίηση είναι απαραίτητη ακριβώς για να εντοπίσουμε τι συμβαίνει στον έξω κόσμο και πώς αλλάζουν οι μεταναστευτικές ροές γενικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καινούριο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η δραστηριότητα ε, ε μόνιμη και online στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι σημαντικό γιατί δίνει και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για να έχουμε μια καλή εικόνα των ε, δυνατοτήτων των κρατών μελών. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο ταυτόχρονα και ε, τι γίνεται εκτός Ένωσης και τι γίνεται εντός και ε, στα κράτη-μέλη μπορούμε να συντονιζόμαστε, να βλέπουμε ποιες είναι οι ισορροπίες κάποια στιγμή και πώς μπορούμε να τις ε, προλάβουμε και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση τους. Ένα τελευταίο, χωρίς αυτό να είναι λιγότερο σημαντικό, εξωτερική διάσταση και η μετεγκατάσταση, η επανεκατάσταση, το resettlement. λόγω ε, και δημοσιονομικών δυσκολιών αλλά και επειδή είμαστε στην αρχή της προσπάθειας αυτής ε, δεν μπορούμε παρά να έχουμε περιορισμένη προσοχή σε αυτό ως βασική υποστήριξη επιμέρους. γιατί έχουμε και ε, πολύ ε, επίγουσες καταστάσεις και πολύ μεγάλες προτεραιότητες. Όπως είπα και προηγουμένως, μία από τις φιλοδοξίες που έχω στην ΕΑΣΟ είναι όχι απλώς να έχουμε μια πρακτική συνεργασία και να παρέχουμε υποστήριξη στα κράτη-μέλη, αλλά να έχουμε και ε, πληροφόρηση τεκμηριωμένη βάσει στοιχείων και από τη βάση προς την κορυφή. Καταφέραμε να το κάνουμε αυτό πέρσι ήδη σε δύο σημεία και σε δύο φάσεις, την έγκαιρη προειδοποίηση με την ενημέρωση και με την πραγματογνωμοσύνη που έχουμε και την εμπειρία. Μέχρι τώρα καταφέραμε να ε, δώσουμε ε, στους πολιτικούς ε, την εμπειρία μας και ελπίζω να έχουμε συνεισφέρει και για τον κανονισμό Δουβλίνο 2 στην τελική του μορφή. Για τη μετακατάσταση τώρα ή την επανεκατάσταση είναι ένα ε, ζήτημα άκρος πολιτικό. Έχω πλήρη επίγνωση αυτού και καταφέραμε να δούμε τα σχέδια Γιουρίμα 1, Γιουρίμα 2 και τα διμερεί σχέδια μεταξύ των κρατών μελών και της Μάλτας και ε, εξάγουμε τις εμπειρίες, τα συμπεράσματα και τα στοιχεία που μας χρειάζονται. Με αριθμούς και ε, στοιχεία που θα συγκεντρωθούν σε μία έκθεση. Και πάλι ε, από τη βάση προς την κορυφή, από τις επιτόπου πληροφορίες. Για να ολοκληρώνω, Πρόεδρε, η διαδικασία λοιπόν έναρξης των εργασιών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά εργαζόμαστε πλήρως ήδη για τις περισσότερες ε, εργασίες που καθορίζονται στον κανονισμό. Έχουμε κάνει ε, βήματα πρόοδου και για τα μεμονωμένα έργα και τα μεμονωμένα σχέδια σε συγκεκριμένες περιοχές. Όπως είπαμε είναι κατάρτιση, εκπαίδευση και αυτό νομίζω τώρα εδραιώνεται ως ε, οργανωτικό σχήμα μέχρι στιγμής. Αυτό πρέπει να το κάνω σε συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και το κατανοώ και κάνω ό,τι μπορώ για να συμμορφώνομαι. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιτροπή σας για την υποστήριξή σας στη δημοσιονομική για τις τροπολογίες που ψηφίσατε. Κρίμα που δυστυχώς δεν εγκρίθηκαν ε, πλήρως ε, τελικά στο βαθμό που θα επιθυμούσε κανείς, αλλά αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από πλευράς της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ταυτόχρονα, επειδή βλέπουμε λοιπόν να περιορίζεται ο προπολογισμό μας, θα καταλάβετε κι εσείς ότι πρέπει να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες. Γι' αυτό τι σημαίνει ότι και το 2013 η ΕΑΣΟ δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από τον κανονισμό. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κρίμα ε, και δεν με ικανοποιεί καθόλου, αλλά... Νομίζω ότι είναι ισόρροπη η επιλογή που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και ακριβώς όταν επήγουν κάποιες καταστάσεις επήγει και να δοθεί προσοχή. Ευχαριστώ κύριε Βίσερ. Πριν δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιος αρμόδιος ε, έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνεργαζόμαστε συνεχώς και πολύ στενά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΑΣΟ. Ε, οπότε, ε, βεβαίως, ε, προσυπογράφουμε και την ετήσια έκθεση και ευχαριστούμε Ε, όπως συμβαίνει πάντα με τις εκθέσεις, υπάρχει χώρος για βελτίωση και θα συνεργαστούμε για τη δεύτερη εκδοχή της έκθεσης που θα ε, εκδοθεί του χρόνου. Θα ήθελα να τονίσω εγώ ένα σημαντικό στοιχείο που έχουμε ήδη συζητήσει με την ΕΑΣΟ για να βρούμε μια λειτουργική λύση και να συντονίσουμε του χρόνου την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ετήσια έκθεση του ΕΑΣΟ για να ε, έχουμε ένα μήνυμα ενιαίο για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και λεπτό όπως είναι το άσυλο. Αυτή ε, εγκρίθηκε από την, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΟ για να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των δύο εκθέσεων του χρόνου λοιπόν. Και μια που αναφερθήκατε ήδη ε, στο 2013, θα ήθελα να σας πω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιάσο, θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο για τη συνεκτική εφαρμογή του νέου κεκτημένου για το άσυλο, ως προς την κατάρτιση και την εκπαίδευση και την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών ενημέρωση με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Και καλό θα ήταν και για να πετύχει το νέο σύστημα ασύλου έχει κομβικό ρόλο να διαδραματίσει άσο και με τα κράτη-μέλη στη συνεργασία αλλά και κάτι άλλο τα επόμενα έτη η ΕΣΟ θα δίνει σημαντική πληροφόρηση για να υπάρχει και ε, συνεκτική και αποτελεσματική παρακολούθηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχουν τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Μπουσουτήλ πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΑΣΟ. Θα ήθελα καταρχάς να τον ε, συγχαρώ για την εργασία του. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιήθηκε για την προώθηση του κανονισμού που συντάχθηκε στην υπηρεσία σας. Χαίρομαι τώρα που μεταφερθήκατε στο νέο κτίριο. Δεν είχα μέχρι τώρα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην εναρκτήρια τελετή, αλλά σας συγχαίρω που μεταφερθήκατε, εν πάση περιπτώσει, στην καινούργια σας έδρα και τώρα μπορείτε πλέον με την αναγκαία υποδομή να λειτουργήσετε πλήρως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο σας και από την ε, πλευρά του προϋπολογισμού. Αναφέρετε την έννοια λιτότητα βεβαίως, αλλά η Επιτροπή μας έχει δηλώσει σαφέστατα ότι θέλει να υποστηρίξει την υπηρεσία σας με όλα τα κονδύλια, με όλες τις πιστώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή έτσι ώστε η, το ΕΑΣΟ να μπορέσει να αποδώσει όπως χρειάζεται. Η έκθεση Τριανταφυλλίδη έχει υιοθετηθεί αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Είναι μία ε, πρωτοπόρος έξεση η οποία εκπροσωπεί τις απόψεις του σώματος εδώ και πολλά χρόνια, αλλά παρουσιάζει και συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση του ζητήματος. Αναφέρεται συγκεκριμένα στην υποστήριξη της επανεγκατές της επανεγκατάστασης και τα πλεονεκτήματα ε, της διεθνούς συνεργασίας και θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, κύριε Ρευθυντά, το άρθρο 5 του κανονισμού σας αναφέρει ότι είσαστε υπεύθυνο, έχετε μία σαφή ευθύνη για την υποστήριξη και μάλιστα την προώθηση, τη διευκόλυνση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την επανεγκατάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα σαφές καθήκον το οποίο έχει η υπηρεσία σα και αναμένω από την ΙΑΣΟ να αναλάβει την πρόθεση διευκόλυνση το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την επανεγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι ιδιαίτερα που πολύ περιορισμένη συζήτηση έχει γίνει από αυτού του θέματος, ακόμα και μέσα στην ΕΑΣΟ και ελπίζω να μπορέσει να αναλάβει από μόνο της πρωτοβουλίες και να μην περιμένει ούτε από την Κομισιόν ούτε από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν μόνα τους. Εάν περιμένουμε από τους άλλους, από τα κράτη-μέλη και να, να αναλάβουν αυτή την ε, δραστηριότητα δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει από το 2009 ότι υποστηρίζει έναν μόνιμο μηχανισμό επανεγκατάστασης και ακόμα δεν έχουμε δει τη συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι. Στο άρθρο 5 όμως του κανονισμού δηλώνει σαφέστατα και δεσμεύει την ε, Κομισιόν όσον αφορά ε, την υπηρεσία, όσον αφορά την προώθηση, το συντονισμό ε, της επανεγκατάστασης. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται για την υλοποίηση του άρθρου 5. Ο κύριος Η κυρία Ρομέρο. Η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω κύριε για την ενημέρωση. Κρίμα που τα έγραφα μας ήρθαν σήμερα και δεν μπορέσαμε να τα διαβάσουμε. Και δεν επεκταθήκατε εσείς πάρα πολύ ε, ως προς τα συμπεράσματα που θα θέλετε να μας διαβιβάσετε Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς ε, ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση για να τροποποιηθεί ο κανονισμός Δουβλίνο 2. Γιατί όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Μπουσούτηλα, εσείς έχετε αυτή την ευθύνη από τον κανονισμό και επιθυμούμε να μας πείτε τι λύση προτείνεται να δοθεί σε όλες αυτές τις χιλιάδες ετούντες άσυλο που δεν έχει λυθεί η κατάστασή τους ούτε στη Μάλτα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Ε, από όπου έχουμε, πει, ε, έχουμε δει, δει σώμαση με τις επισκέψεις μας οι βουλευτές. Πρόσφατα είχαμε μια αποστολή στην Ελλάδα και η Άσο εκεί εκπροσωπείται από έναν υπάλληλο. Έτσι μας είπε ο υπάλληλο και ο εκπρόσωπός σας στην Ελλάδα. Το ξέρω ότι υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε σύστημα ασύλου με τέτοια χρηματοδότηση. Σε εμάς εναπόκειται βεβαίως ε, αυτό το έργο και έχουμε αφιερώσει και όλο τον προϋπολογισμό εκεί ε, μόνο σε κατασταλτικά μέτρα, αποκλειστικά. Άρα είναι προφανές ότι η υπηρεσία ασύλου και το σύστημα ασύλου κοστίζει χρήματα. Και αν δεν κοστίζει εκεί χρήματα, κοστίζει αλλού, στην καταστολή και σε άλλε καταστάσει που θα ήταν πολύ λιγότερο επιθυμητέ. Θα ήθελα να μιλήσω βέβαια και να μα μιλήσετε και για τα κέντρα κράτηση, γιατί έχετε και ευθύνη να ε, κρούετε τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση εκεί που επικρατεί. Δεν μπορούν να κάθονται οι άνθρωποι τρει και έξι μήνες ε, σε ε, συνθήκες που δεν είναι αντίστοιχε της ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν είναι εγκληματίε, αλλά και εγκληματίε να ήταν. Είδαμε κέντρα κράτησης με συνθήκες ικτρές, πώς να το πω. Ζητήσαμε στην Ελλάδα να κλείσουν δύο κέντρα, στη Βένα και στο Παλιό Ελληνικό. Δύο κέντρα κράτησης εκεί, δύο κρατητήρια. Προσωπικά έχω πάει και σε άλλα. Και σε άλλες χώρες θα πρέπει να κλείσουν άλλα κέντρα. Βεβαίως χρειάζεται να δράσει εκεί η ΕΑΣΟ, διότι τα κράτη-μέλη κανονικά θα πρέπει να δουν, να διαμαρτυρηθεί κάποιος. Τι γίνεται με την κατάσταση αυτή στο άσυλο, δεν απαντούν. Στην Ελλάδα δεν ξέρουν και πόσες είναι οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν. 50.000, 25.000. Και με το νέο νόμο για το άσυλο στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν ακόμα σε ποιο αριθμό θα καταλήξουν. Και δεν μπορούμε να αφήνουμε χρόνια ολόκληρα άνθρωπους που έχουν ζητήσει άσυλο χωρίς ε, απάντηση. Είναι προτεραιότητα αυτή η προσέγγιση. Για μας τους βουλευτές εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να είναι προτεραιότητα. Στην Ελλάδα τώρα εστιάζει ε, η ΕΑΣΟ. Σωστά, έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική ασύλου χωρίς να λησμονούμε και την ε, εξωτερική πολιτική και τις δικές μας ευθύνες και εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, παρευρίσκονται. Αλλά αν δεν το δούμε ολοκληρωμένα και συνολικά είναι σημαντικό το θέμα. Υπάρχει και το θέμα των πρεσβειών και πώς συνεργάζονται οι χώρες και οι πρεσβείες. Τα γνωρίζετε κι εσείς αυτά τα θέματα. Χρειάζονται ε, αυτοί οι άνθρωποι κάποια χαρτιά από τις πρεσβείες τους, ε, ε, βασικά έγγραφα, ένα λεσέπασε και όλα αυτά καθυστερούν και έχουμε αλληγορίες γιατί δεν θεωρήθηκε το θέμα προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν μπορούμε να έχουμε χιλιάδες ανθρώπους σε τέτοια κατάσταση που ζουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο. Κυρία Βίξτρομ. Και βιαστείτε, 9 και 45 έχουμε μακρά ακρόαση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Με τρεις ε, στρογγυλές τράπεζες και τα λοιπά. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Βίσερ για την παρουσίαση και για το πρόγραμμα το οποίο μας στείλετε μέσω του, ε, του ίντερνετ. Επειδή είμαι και η συγγήτρια για το Δουβλίνο 2, θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου για το άρθρο 31 πιο συγκεκριμένα, το οποίο θίξετε και εσείς στην ε, παρέμβασή σας. Όπως ξέρετε, το άρθρο 31 αναφέρεται σε έναν έγκαιρο μηχανισμό ε, προειδοποίησης μέσα στα πλαίσια του Δουβλίνου 2, έτσι ώστε να ε, βρεθούν τα προβλήματα στα εθνικά συστήματα ασύλου πριν τα προβλήματα αυτά ε, μετατραπούν σε κρίσεις. Αυτό είναι το εργαλείο μας επομένως για να αποφύγουμε ε, να εμφανιστεί μια άλλη περίπτωση έκτακτης ανάγκης σαν και αυτή της Ελλάδας, όπου εκεί το σύστημα κατέρευσε και υπάρχουν κάποιοι ρόλοι κλειδιά που ε, δηλαδή σε ε, φορείς που πρέπει να στην ΕΑΣΟ που πρέπει να παρακολουθούν και να ε, αντιδράσουν. εστιάστηκαν, εστιάστηκε πολλές φορές η ΆΣΟ στα κράτη-μέλη σε, περίπτωση, σε περιπτώσεις προβλημάτων, όμως θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα κράτη-μέλη και όχι μονάχα τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες πιέσεις, όχι μόνο δηλαδή τα κράτη μελη της Νοτίου Μεσογείου, γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη. Και εφόσον το σύστημα του Δουβλίνου στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι το σύστημα ασύλου θα πρέπει να προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις σε όλους όσους, ετούνται άσυλο, χρειαζόμαστε μια πολύ προσεκτική παρακολούθηση όλων των κρατών μελών. Επίσης, στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΣΟ για το 2013 διαβάζουμε την πρόθεσή σας για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ρωτώ, θεωρείτε ότι έχετε επαρκείς πόρους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους έτσι ώστε να καλύψετε αυτά τα τεράστια καθήκοντα τα οποία σας έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 31, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που αντιμετωπίζουμε και τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Επίσης ε, θα ήθελα να μας πείτε λίγα περισσότερα για την δυνατότητα ελέγχου όλων των κρατών μελών και όχι μόνο αυτών που βρίσκονται στα νότια σύνορά μας, στη Μεσόγειο και θα ήθελα να μας πείτε εάν προβλέπετε κάποια προβλήματα με την θέληση των κρατών μελών να συνεργαστούν και τι, για να σας δώσουν και τα στοιχεία τα οποία ζητείτε εσείς αλλά και να εφαρμόσουν τα συστήματα, τους μηχανισμούς πρόβληψης που ε, προτείνετε εσείς ή τι άλλο τέλος πάντων ε, ε, ζητάτε. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον κύριο Βίσερ για την ομιλία του και ε, επίσης και για όσα κάνει το γραφείο του για τους ετούντες άσυλο. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τα γραφεία στην Μάλτα και συζήτησα πάρα πολύ ε, ωραία με τον διευθυντή εκεί και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένο ε, με την δουλειά που κάνω, διότι έχω δει τα αποτελέσματα της δουλειάς τους ε, όταν επισκέφθηκα και την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Όμως θεωρώ ότι και οι ελληνικές αρχές είναι ικανοποιημένες διότι έχουν την άμεση βοήθεια της ΕΑΣΟ, της ΕΑΣΟ για, να κάνουν, για να εφαρμόσουν αυτές τις τόσο σημαντικές πολιτικές στον τομέα του ασύλου. Και προφανώς περιμένουν και πολύ περισσότερη βοήθεια για την ε, ε, θέσπιση και εφαρμογή των ε, νέων υπηρεσιών για το άσυλο που ναι, ναι, ναι είναι έτοιμη σχεδόν, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα όμως. Μία ερώτηση που την έθεσε και ένας συνάδελφος για την επανεγκατάσταση. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιό κατά πόσον προτίθεται να υποβάλει μία πρόταση για το θέμα αυτό και για τα κατά πόσον θα υπάρχει μία θεσμική κλίδα κατανομής. Επίσης, ε, το, η αξιολόγηση του προγράμματος Γιουρίμα, του Γιουρίμα 2. Πώς θα προχωρήσει αυτό για το θέμα, στο θέμα αυτό. Επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση που έγινε για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. η χώρα προέλευσης, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις ε, ε, χώρες, να, τις αρχές να αποφασίσουν για την αίτηση ασύλου και κατά πόσο να ε, προβλέπουν να έχουν πρακτικά αποτελέσματα. Ο κύριος Κάποιε ερωτήσει, Κάποιες ερωτήσεις και ε, τις οποίες έχω θέσει και σε άλλου στο παρελθόν, αλλά δεν έχω πάρει καμία ικανοποιητική απάντηση. Ποιο είναι το ποσοστό των ετούντων άσυλο έχουν ε, επιλεγεί για την, ε, για τις, από τις λόγω των, της χώρας ε, προέλευσης ή, και πόσοι αιτούνται σε άσυλο έχουν, τους έχουν αρνηθεί γιατί θεωρούν ότι είναι επικίνδυνοι τον πληθυσμό. Επίσης, πιο συγκεκριμένα, ποιο είναι το ποσοστό των αιτούντων άσυλο που δεν τους χορηγείται τελικά άσυλο. Επίσης, ελέγχεται ο αριθμός... αυτών που, τους οποίους έχει αρνηθεί, τους έχουμε αρνηθεί την αίτηση κατά πόσον επιστρέφουν ε, στη χώρα τους. Η Frontex, ο διευθυντής της μας είπε ότι και οι παράνομοι μετανάστες και αυτοί οι οποίοι ζητούν ε, άσυλο και δεν τους δίδεται, δεν ε, απομακρύνονται, τους δίδεται όμως μια εντολή απομάκρυνσης που όμως δεν εκτελείται. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν χτες είπε ότι υπήρχε μία μετακίνηση από την υποχρεωτική απομάκρυνση στην προαιρετική απομάκρυνση ή εθελούσια απομάκρυνση. Ρωτώ, έχετε ένα ανώτατο όριο στους ετούντες άσυλο που στην Ευρώπη ή θα είναι ο αριθμός ε, χωρίς κανένα όριο. Επίσης, με ανησυχεί ο αριθμός των ετούντων άσυλο που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχει, υπάρχουν συγκρούσεις, πολεμικές εχθροπραξίες και που ε, ενθαρρύνονται από δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πιο συγκεκριμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, ανησυχώ πολύ διότι χώρες που τώρα έχουν επιστρέψει φαίνεται στην δημοκρατία έχουν ε, εδώ ε, σαν σύλλο. Ας πούμε, την Ίση ε, προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα τους λόγω του προηγούμενου καθεστώτας. Τώρα όμως που υποτίθεται ότι τα πράγματα έχουν επανέλθει στην, στο κανονικό τους, αυτοί την ίση δεν θέλουν να επιστρέψουν. Ευχαριστώ. Κύριος Βίσερ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω ε, ανατομής και θέμα της ερωτήσης. Ίσως είναι πιο πρακτικό αυτό. Καταρχάς θα ήθελα και πάλι να σας εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη της Επιτροπής σας, στο σύνολό της. Αλλά και βουλευτές ε, μεμονωμένα ε, έδειξαν ε, προς την ΕΑΣΟ επανειλημμένα δέχτην πρόσφατα την επίσκεψη ε, στη Μάλτα πολλών από εσά και αυτό είναι ε, μήνυμα θετικής υποστήριξης πάρα πολύ σημαντικό για ε, μια νέα υπηρεσία. Για τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Ίσως να ξεκινήσω από την ετήσια έκθεση που είναι το θέμα στην ημερήσια διάταξη που μας απασχολεί. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε τώρα, ούτε μπήκα προηγουμένω γιατί δεν είχαμε χρόνο, ε, λόγω και του χρόνου που μου έδωσε ο πρόεδρο. Δύο λόγια μόνο. Είναι η πρώτη ετήσια έκθεση. Ε, συνδυάζουμε ουσιαστικά εδώ δύο εκθέσει. Η μία είναι η έκθεση για την κατάσταση προ το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο είναι η έκθεση πεπραγμένων ή ε, δραστηριοτήτων μα. Ε, του χρόνου θα διαχωρίσουμε τις δύο εκθέσεις και θα έχουμε την έκθεση δραστηριοτήτων ξεχωριστή ε, ως λογοδοσία για τον προϋπολογισμό και ε, θα κάνουμε μια χωριστή έκθεση πλέον για την κατάσταση ε, ως προς το άσυλο στην Ένωση του χρόνου, επαναλαμβάνω. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς επίσης να έχουμε και μια συνολικότερη ε, εικόνα και επισκόπηση για το τι συμβαίνει στον τομέα του ασύλου. Όπως είπε ήδη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε επικαλύψεις και ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση γενικά ε, θα εγγράφεται στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια σειρά, η Λουχία μάλλον εμεί θα ακολουθούμε τη σειρά της ευρύτερη εκθέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ε, άλλε εκθέσεις όπως αυτές της Eurostat και θα έχουμε στενό συντονισμό. Αυτά είναι τα διαδικαστικά για τις εκθέσεις. Στη συνέχεια, και πάρα πολύ σημαντικό, το 2013 θα είναι το λεγόμενο πακέτο ασύλου, που βεβαίως θα πρέπει να κυρωθεί από όλους τους ενεχομένους και ε, όπως έχει η κατάσταση των πραγμάτων σήμερα μπορούμε να προβλέψουμε ότι για σημαντικά θέματα ε, ήδη από το 2013 το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα αλλάξει και θα βελτιωθεί. Αυτό τι σημαίνει. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει τα επόμενα έτη να εφαρμόσουν νέα νομοθεσία αλλά και νέες πρακτικές για το άσυλο. Και αυτό αγγίζει πλέον και τον πυρήνα των καθηκόντων ε, της υπηρεσίας μας, να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, ε, να διοργανώσουμε, ε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην οργάνωσή τους, στην βελτίωση της ποιότητας σε αυτή τη διαδικασία και δεδομένου του προϋπολογισμού και των προτεραιοτήτων. Βεβαίως αυτό το λεγόμενο πακέτο για το άσυλο του 2012 θα είναι πολύ σημαντικό, κλειδί θα έλεγα, για να δούμε πού θα μπουν οι προτεραιότητες για την επόμενη διετία. Τρίτο θέμα, η επανεκατάσταση. Σωστά αναφερθήκατε σε αυτό. Ο κύριος Μπουσουτήλ και κάποιοι άλλοι βουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό. Μα γι' αυτό άλλωστε αναλάβαμε και την πρωτοβουλία. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανεξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τη Γιουρίμα 1, Γιουρίμα 2 και τα συστήματα διμερής υποστήριξης της Μάλτας. Διμερούς υποστήριξης. Ε, στα μέσα του έτους είχαμε και εκθέσεις ε, μετά από επισκέψεις επιτόπου και στο Λουξεμβούργο πριν από 10 μέρες συζητήθηκε αυτό το θέμα σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια και θα παρακολουθήσει το θέμα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δική μας δράση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί έχουμε ήδη δράσει σε αυτό το τομέα, θα συμμορφωθούμε πλήρως στον κανονισμό, θα προωθήσουμε και θα διευκολύνουμε τη διαδικασία πανεγκατάστασης όταν αυτή συμβαίνει. Ταυτόχρονα ε, οφείλω να πω και το εξής και προς τον αξιότιμο κύριο Μπουσουτήλ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα πολιτικά φορτισμένο. Και η ε ΕΑΣΟ και ο κανονισμός της ΕΑΣΟ ορίζει ότι συντονίζει, αλλά δεν μπορεί να αναλαβεί την πρωτοβουλία ή την ηγεσία σε αυτή την προσπάθεια η ΕΑΣΟ. Έχω δει ήδη αρκετές ε, δυνατότητες, ε, κινώντας από τη δική μας αξιολόγηση, για να διαδραματίσουμε σωστά το ρόλο μας και είδα αποδοχή από τα κράτη-μέλη για το ρόλο τον οποίο παίζουμε. Τώρα αναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση ε, μετά από τις συζητήσει σε πολιτικό επαναλαμβάνω επίπεδο και ταυτόχρονα και παράλληλα η ΆΣΟ θα συνεχίσει να οργανώνεται και με τα δικά της μέσα και το ρόλο της να παίζει στην επανεγκατάσταση. Δεν θα είναι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο όμως ε, στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση. Ελλάδα. Ακούστηκαν πολλά ζητήματα εδώ σχετικά με την Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Ο κανονισμός ορίζει ότι η ΆΣΟ ε, μπορεί να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη μόνο κατόπιν ρητού αιτήματο του συγκεκριμένου κράτους. Έχει γίνει αυτό με την Ελλάδα και Έχουμε υποστηρίξει μέχρι τώρα την Ελλάδα σε όλες τις δραστηριότητες και σε όλες τις δράσεις όπου θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην οργάνωσή τους. Τώρα είμαστε μια πλήρως τελεχωμένη υπηρεσία και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ε, ε, τους Έλληνες για να στήσουν τις τρεις ε, νέες, τρεις δομές για το άσυλο. Υπό την προϋπόθεση ότι ε, η στελέχωση και η οικονομική πόρη είναι δεδομένη ε, από την ελληνική πλευρά. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Γι' αυτό δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι δομές αυτές, οι υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αλλά μόλις στελεχωθούν και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, ε, είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα έχουμε εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό των υπηρεσιών, τους έχουμε υποστηρίξει και διοικητικά, τους έχουμε δώσει εγχειρίδια, κατευθυντήριε γραμμέ, εσωτερικές εντολές για ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη κατάρτιση για βάλετες ομάδες, ασυνόδευτους ανηλίκους, διαχείριση και διοίκηση κέντρων υποδοχής. Οι νέες υπηρεσίες είναι λοιπόν έτοιμες, είναι κατερτισμένε ε, και σε καλό επίπεδο έχουν προχωρήσει οι εργασίες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα ε, πέρα από τη μετάβαση είναι ε, η ε, συσσόρευση, η καθυστέρηση στις αιτήσεις ασύλου, το λεγόμενο backlog. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό για τις νέες υπηρεσίες να μην έχουν όλη αυτή τη βαριά κληρονομιά. Γι' αυτό Συνεργαζόμαστε με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Έχουμε ένα κοινό έργο και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να αποφασιστεί και να καταλήξει αυτό για να προχωρήσουμε σε ένα έργο που θα επικεντρωθεί ε, στην ε, αντιμετώπιση αυτής, αυτού του όγκου που έχει συσσωρευτεί. Να βοηθήσουμε την Ελλάδα με το νέο σύστημα ασύλου ε, που αρχίζει τώρα. Λοιπόν, για την έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το άρθρο 31 η Άσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζουν εδώ ρόλο κλειδί. Η Άσο στη φάση ε, της ε, δημιουργίας της εικόνας, ας πούμε, της εκτίμησης, της παρακολούθησης για το πώς έχει η κατάσταση. Λίγα ε, συγκεκριμένα να σας πω. Συμφωνώ τους ότι θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία, διότι εάν θέλετε να είστε ε, προετοιμασμένη γιατί αυτό είναι η εγκαιρή προειδοποίηση. Δεν είναι ένα σύστημα ε, τιμωρίας, δεν είναι το πρώτο βήμα προς την προσφυγή επί Όχι, είναι προειδοποίηση για να μπορεί να προετοιμαστεί το κράτος, όχι να του επιβάλλουμε κάποια κύρωση. Ένα ειδικό παράδειγμα. Αρχές του έτους πήρε ένα σήμα προειδοποιητικό. Το Λουξεμβούργο, άκουσαν, άκουσαν, το Λουξεμβούργο. Δεν θα το περίμενε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Αλλά το Λουξεμβούργο είχε μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι θέμα Μεσογείου, δεν είναι θέμα ανατολικών συνόρων, είναι για όλα τα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια και ναι και όχι. Δεν είναι δύσκολη διότι οι πάντες κατανοούν ότι χρειάζεται συνεργασία για να καταλάβουμε πώς έχει η κατάσταση και ποια είναι η εικόνα. Και η εικόνα μπορεί να είναι κάτι που αφορά το γείτονά σου. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοιχτά σύνορα. Αυτό που συμβαίνει στο γείτονα μπορεί να σε επηρεάσει άμεσα. Οπότε, εάν δεν συνεργάζονται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όλοι, δεν θα δουλέψει. Το θέμα δεν είναι μόνο η πληροφορία, είναι να βάλει ο καθένας ε, το λιθαράκι του για να βγει το ψηφιδωτό σωστό. Ξέρω ότι αυτό είναι υποσυζήτηση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορούμε να στήσουμε το σύστημα. Εργαζόμαστε, ε, αφιερώνουμε πόρους και ανθρωπινούς και οικονομικούς, αλλά αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ έντονη. Ξέρετε, αν θέλετε πραγματικά να ελέγξετε την κατάσταση στα κράτη-μέλη με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε, όχι βέβαια να προβλέπετε, είναι πολύ βαριά λέξη η πρόβλεψη, αλλά να δίνετε μία ένδειξη, με ανάλυση κινδύνου, ανάλυση κάποιων τάσεων ε, με τρόπο έτσι που να ευσταθεί, ε, χρειάζεστε ε, προσωπικό εξειδικευμένο. Εδώ είναι πιο σημαντική η ανθρώπινη πόρη παρά η οικονομική αυτή καθ' αυτή. Θα πρέπει να έχουμε αφοσιωμένο προσωπικό και καλά κατηρτισμένο. Λοιπόν, ίσως χρειαστεί να επανέλθω σε αυτό όταν θα έχουμε περισσότερη εμπειρία. Βλέπω τον Πρόεδρο. Ναι, ξέρετε, έχουμε ακρόαση, γιατί πρέπει να έχει αρχίσει από τις παρατέταρτο. Uh, Τότε, καταλήγοντας, να αναφέρω ένα θέμα μόνο, ένα σημείο, την, τη διάσταση του ασύλου, εάν υπάρχει ένα ανώτατο όριο στους ετούντες ασυλό οι αξίες τις οποίες όλοι πιστεύουμε λένε ότι μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν όρια στην, στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στο να φανούμε άνθρωποι στους άλλους. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισήγησή σας και για τις προσεκτικές απαντήσεις σας και σας ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν σύντομος δεδομένου ότι βρισκόμαστε υποπίεση χρόνου ε, ευθύ εξ αρχή. Διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε, θα έπρεπε να είχαμε αρχίσει δηλαδή, ε, την ακρόαση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ελπίζω να σα ξαναδώ σύντομα. Yes. Good morning. So, no further delay. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση, δεδομένου ότι όπως σας είπα ήδη έχουμε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα που πρέπει να εκτελέσουμε. Έχουμε 2 ώρες και 15 λεπτά να ε, εξετάσουμε ακριβώς, να κάνουμε αυτή την ακρόαση. Και θα ήθελα να σας πω ακριβώς ποια είναι αυτή η βασική ιδέα. Uh, uh, Γι' αυτό λοιπόν οι εργασίες της Επιτροπής μας, ΛΥΜΠΕ, έχει υποβάλει την έκθεση για το ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο θα θέτει τα, τους κανονισμούς για την ε, ελευθερία του τύπου η συγγήτρια Ρενάτε Βέμπερ ε, ε, Άλντε και γι' αυτό οργανώσαμε ακριβώς αυτήν την ακρόαση και την συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους για να τονίσουμε ακριβώς την έκθεση αυτή η οποία θα έρθει στα χέρια μας σύντομα. Παρακαλώ πολύ να είστε ησυχία. Ο πρόεδρο ζητά ησυχία από τους ε, ακροατέ, διότι πρέπει να διεξάγουμε την ακρόαση. Παρακαλώ ησυχία. Και... Ε, όσοι είσαστε στην αίθουσα και περιδιαβάζετε, παρακαλώ αποχωρήστε, διότι θέλουμε να αρχίσουμε τι εργασίε μας με την ημερήσια διάταξη καταρχάς. Ε, η οποία οργανώθηκε από τη συνάδελφό μας την Ρενάτε Βέμπερ. Έχουμε λοιπόν τρεις εισηγήσει κάθε μία θα, μετά από κάθε μία θα ακολουθήσει συζήτηση, θα καταγράψουμε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις και προτείνω δεδομένου ότι έχουμε 2 ώρες 15 λεπτά διότι στις 12.30 πρέπει να ολοκληρώσουμε διότι έχει, έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Λοιπόν, 12.30 ώρα ακριβώς πρέπει να τελειώσουμε. Το πρώτο πάνελ λοιπόν μας θα ξεκινήσει με τη συνάδελφό μας κυρία Βέμπερ και έχουμε τρεις καλεσμένους. Την κυρία Λεωνόρα Γαβριλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Είναι η Διευθύντρια του, ταμείου, του Γραφείου ε, Τύπου και Πληροφοριών της, της ε, Κυπριακής Προεδρίας. Για συνεχεία έχουμε τον κύριο Άντωνη Βίλαν, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου της ε, κυρίας Νέλη Κρός, η οποία είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή ατζέντα και την κυρία Ντάντζα Μιλιάτοβιτς ε, από πλευρά ΟΑΣΕ. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ρενάτε Βέμπερ, η οποία προεδρεύει του πρώτου πάνελ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους όσοι είναι παρόντες σήμερα. Θέλουμε σήμερα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και να βοηθήσουμε τους νομοθέτες να βρουν τις καλύτερες δυνατόν λύσεις. Όταν θα αποφασίσουν ή όποτε αποφασίζουν ε, για την έκθεση αυτή και γενικά για τα πρότυπα της ελευθερίας του τύπου στην Ευρώπη. θα μιλήσω έτσι καλλιώς για την έκθεση αυτή, θα μιλήσω και για τις τροπολογίες. Απλό, αυτό που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να εξηγήσω γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση πρέπει να ε, παρουσιαστεί το 2012. Ε, μετά από πολλές πρωτοβουλίες και συστάσεις ευρωπαϊκές, ε, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πιστεύουμε ότι όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια τα, πρόβλημα, τα προβλήματα του τύπου ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι του τύπου, τα μέσα ενημέρωση κτλ. μοιάζουν, έχουν πολλές ομοιότητες στα κράτη-μέλη. Και πιστεύουμε ότι ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πολύ σκληρά για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κομισιόν <laughs> είναι μάλλον πολύ συγκρατημένη στο να κάνει κάτι παρόμοιο για πολλούς λόγους. Πολύ συγκρατημένη. Η ιδέα μας λοιπόν ήταν να συντάξουμε μία έκθεση που θα περιλαμβάνει μία δέσμη προτύπων και συστάσεων ώστε να δώσει τη δυνατότητα και στην Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή να υποστηρίξει, να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια δεδομένου ότι είχαμε συγκεκριμένες αναφορές ε, για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το πιο ε, δυνατό, το πιο ισχυρό εργαλείο, το πιο ισχυρό μέσο και πιο ισχυρές διατάξεις που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση σε διεθνές επίπεδο. Εφόσον λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, γιατί δεν έχουμε μια καλύτερη εναρμονισμένη πολιτική ε, μέσω της οποίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις όταν τα μέσα ενημέρωση υφίστανται επιθέσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, βλέπουμε καταχρήσεις, επιθέσεις ε, και παραβιάσεις η έξεση δεν έχει στόχο να εκθέσει και να ντροπιάσει τους ενόχους, αλλά να ε, παρουσιάσει δέσμη κανόνων βάσει των οποίων μπορούν τα κράτη να κρίνουν τι πρέπει να κάνουν ή καλύτερα να ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν. Επίσης ε, υπάρχουν πάρα πολλές αντιφατικές απόψεις, αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό ακριβώς Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τους εκπροσώπους, τους εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Κομισιόν ε, και ταυτόχρονα και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Αυτό ακριβώ είναι ο στόχος της ακρόσης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Και ας ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη ομιλήτρια. Η κυρία Ελεονόρα Γαβριλίδη, Διευθύντρια Επικοινωνιών της Κυπριακ... Επικοινωνίας της Κυπριακής Προεδρίας, έχει το λόγο και Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι αξιωματικό ότι τα μέσα ενημέρωση ε, πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία και είναι δίκαιο να πούμε ότι η ελευθερία αυτή είναι μια προϋπόθεση ύπαρξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τα μέσα ενημέρωση έχουν χαρακτηριστεί ως τέταρτη εξουσία και ο ρόλος τους είναι να προστατεύσει τους πολίτες εναντίον αυθαίρετων και ζημιογόνων δράσεων από τις άλλες τρεις εξουσίες. Βεβαίως υπάρχουν ε, δύο πλευρές στο νόμισμα και πολλές φορές οι κυβερνήσεις πρέπει να προφυλαχθούν έναντι αντιδημοκρατικών πρακτικών. Πράγματι, τα μέσα ενημέρωσης μπορεί πολλές φορές να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να έχουν μεγάλη επιρροή. Στην Ευρώπη είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε καθιερώσει τη δυνατότητα ελευθερίας έκφρασης, ελευθεροτυπία και δικαιώματα τα οποία έχουν χαραχθεί, έχουν ε, ε, καλυφθεί από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αυτομάτως υλοποιούνται και εφαρμόζονται ή υλοποιούνται με τον τρόπο που αρχικά είχαμε επιδιώξει. Ό, σημαίνει όμως ότι τα κρατη και τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη όργανα έχουν ένα πολύ δυνατό ε, εργαλείο στα χέρια της για να εφαρμόσουν ακριβώς την ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Είναι γεγονός ότι δεν ζούμε σε έναν παράδεισο. Υπάρχουν πολλά αρνητικά παραδείγματα, βλέπουμε πως αυτή τη στιγμή τον ξεσηκωμό των αραβικών χωρών και πώς ξεκινούν ε, με ένα καινούριο τρόπο αντιμετώπιση της ελευθεροτυπίας και των μέσων ενημέρωσης και πραγματικά μας καθιστά πολύ ταπεινούς η γνώση ότι και εμείς δεν έχουμε φτάσει σε μια ιδανική κατάσταση ακόμα. Αν εξετάσετε την έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ιδίως σε εποχές οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα και η Ιταλία αυτή τη στιγμή έχουν μια πάρα πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 70η και 61η αντίστοιχα. Η Βουλγαρία 80η, η Λουθουανία και η Λετωνία επίσης έχουν πέσει από την 30η στην 50η θέση. Το Ενωμένο Βασίλειο χαμηλά στην 28η, η Γαλλία ακόμα χαμηλότερα στην 38η. Αυτοί οι δείκτες δείχνουν ότι ε, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες ε, μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις όπως παραδείγματο χάρη το σπίτι της ελευθερίας με την έκθεσή του για την ελευθερία του τύπου Προφανώς σε αυτή την έκθεση επίσης η Φιλανδία, ο συνήθως η Νορβηγία, η Ολλανδία, ε, η Ισλανδία, η Αυστρία, η Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Δανία, η ε, Δημοκρατία της Τσεχίας, ε, η Κύπρος και η Γερμανία είναι στις πρώτες 16 χώρες και που λαμβάνουν και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως ο Κανάδας, η Νέα Ισλανδία και, και η Πράσινη Ακτή. Το Κέμπ το πράσινο, το ακροτήριο. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Περισσότερη και πιο συντονισμένη δραστηριότητα εργάζεται, ε, χρειάζεται για να εδραιώσουμε και να διασφαλίσουμε αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει και να βελτιώσουμε την κατάσταση που υπάρχει εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Πολλές φορές βεβαίως ε, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι οι πρώτες χώρες στον κατάλογο αυτό είναι και τόσο ιδανικές, δεδομένου ότι όπως ξέρουμε στη Φιλανδία και στην Νορβηγία, παραδείγματος χάρη, το κράτος επιδοτεί τον τύπο και μπορούμε να θέσουμε νόμιμα το ερώτημα. Είναι σωστό να υποστηρίζει το κράτος ε, τα μέσα ενημέρωσης για να εξασφαλίσει ε, μια ε, πολυμερή διάσταση, ένα πλουραλισμό. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι σωστό. Δεν δημιουργεί όμως και εξάρτηση. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να ξέρουμε τι κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για την ελευθερία του τύπου. Ε, είναι δίκαιο να πούμε ότι η ελευθερία του τύπου διαφέρει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που δίνουν κάποιο είδος επιδότηση ε, στα μέσα ενημέρωση και άλλες χώρες οι οποίες τελείως απορρίπτουν οποιαδήποτε στήριξη και επιδότηση. Γι' αυτό μεταξύ των άλλων έχουν γίνει προσπάθειες για μια διεθνή σύγκριση αυτών των ε, μεθόδων. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ε, ε, ουδέτερα μετρήσιμα στοιχεία και αξιόπιστα, αξιόπιστα δεδομένα. Παραδείγματο χάρη είναι γνωστό ότι οι φοιτητέ τη λογική ξέρουν ότι οι συγκρίσει μπορούν να γίνουν μόνο αν υπά... βάσει συγκρίσιμων δεδομένων. Είναι όμω πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το βρούμε μέσα στο... στον τομέα τη ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωση. Ποιοι τι είναι μετρήσιμο και τι δεν είναι. Υπάρχουν γλωσσικέ διαφορέ, γλωσσικά προσκόμματα, ε, λεπτομέρειε οι οποίε χάνονται όταν κάνουμε συγκρίσει και πολλέ χώρε έχουν μια πολύ συγκεχημένη εικόνα αυτού του τομέα. Γι' αυτό το λόγο όταν εξετάζουμε τις μεθοδολογικές, ε, τις μεθόδους ε, που εφαρμόζονται από τα, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως το σπίτι της ελευθερίας και οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, ε, τα, οι μέθοδοι αυτοί διαφέρουν και χρονικά και τοπικά και πολλές φορές υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την συγκρισιμότητα ε, των στοιχείων και τον κατάλογο αυτό των χωρών που ανέφερα ε, προηγουμένως και την θέση των χωρών σε αυτό τον κατάλογο. Δεν θα επεκτοθώ περαιτέρω σε αυτό, αλλά θα αναφερθώ στις δυσκολίες που υπάρχουν στο κανονιστικό πλαίσιο. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το γεγονός ότι οι κανονισμοί που στοχεύουν στην διασφάλιση της, ε, των διαφορών, της ε, πολυμορφίας, ε, της αποφυγής συγκέντρωσης του τύπου σε λίγα χέρια κλπ πολλές φορές εφαρμόζονται με μέτρα ε, προστατευτικά, κρατικά μέτρα παρέμβασης πειράζει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης η κρατική παρέμβαση ε, θεωρείται ότι ε, συνάδει στην ε, διατήρηση της ποικιλομορφίας. Επίσης τα συμμετοχικά δικαιώματα των δημοσιογράφων. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε σε ορισμένες χώρες. Μέτρα ελευθερίας ερμηνεύονται ως μέτρα περιοριστικά ή επίθεση κατά των δημοσιογράφων. Ήδη έχουμε μιλήσει ότι πολλές μικρότερες χώρες υποστηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης οικονομικά για να εξασφαλίσουν αυτή την ε, πολυφωνία. Αυτές οι αντιθέσεις λοιπόν και αυτές οι δυσκολίες μετρήσεων ε, δεν ε, εκδηλώνται με τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεδομένου όμως ότι αποτελούν ένα σημαντικό δίκτυ των δημοκρατικών αρχών, πρέπει εμείς να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την διαφορά, την ελευθερία του τύπου και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δίκτυ ως δίκτυ ε, μετρήσεως της δημοκρατίας σε οποιαδήποτε χώρα. Να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η ελευθερία των μέσων επικοινωνίας ως δείκτη δημοκρατίας είναι προφανές ότι θα πρέπει να, γίνουν, να δεχθούμε ορισμένες προσαρμογές πολιτιστικές, οι οποίες είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Επίσης, ε, είναι ε, ε, αξιοπρόσεκτο πόσο αποσπασματικές είναι οι προσπάθειες έρευνας οι οποίες γίνεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να επιβάλλουμε ευρωπαϊκά πρότυπα για την ελευθερία του τύπου. Ας ευχηθούμε ότι η διαδικασία της ετήσιας έκθεση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα βοηθήσει τους νομοθέτες ε, στην, ε, στο να ξεπεράσουν ε, τα τεχνικά προσκόμματα. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός ε, Χάρτης ε, σε σχέση με τις, συμβάσει τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ε, ενσωματώσει ακόμα ένα βήμα στο άρθρο 11 παράγραφος 2 προάσπισης της ελευθερίας και του πλουραλισμού. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σήμερα και με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ή δεν θα έχουμε στο, στο μέλλον. Πολλές φορές το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κινείται πάρα πολύ αργά η περιπλοκότητα των συστημάτων μας δημιουργεί καθυστερήσεις. Αλλά αυτό γίνεται επειδή έχουμε πραγματικές δημοκρατίες. Αυτές οι καθυστερήσεις δημιουργούν ορισμένες φορές απογοήτευση ή θυμό, αγανάκτηση. Αλλά αποδεικνύουν ότι εμείς ε, τηρούμε δημοκρατικές μας αρχές και κάθε άλλα αρχή στην οποία η Ένωσή μας βασίζεται. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές είναι καλές, θετικές δυσκολίες, διότι έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ξανά τις καλές μας αρχές τις οποίες πιστεύουμε. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να ε, κρύψουμε το γεγονός ότι πολλά ε, κράτη-μέλη ε, έχουν λήψει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ότι επικρατούν διαφορετικές απόψεις μεταξύ κρατών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να κολλήσουμε στις διαφορετικές ερμηνείες των ορίων ε, της παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να δούμε εάν υπάρχει κάποια νομική ε, βάση παρέμβασης και να επιδιώξουμε μια κεντρική, ένα κεντρικό νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστικό πλαίσιο για την ελευθερία του τύπου εκεί όπου πολιτικά μπορεί αυτό να επιβληθεί και να εφαρμοστεί. Αυτή η συζήτηση έχει τραβήξει πάρα πολύ. Ε, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε συνένεση. Όλοι προσπαθούμε να επιτύχουμε έναν καλό και δίκαιο στόχο. Ας συνεχίσουμε να, τις προσπάθειες αυτές ακόμα και αν κινούμεσα αργά. Θα ήθελα να σταματήσω λοιπόν εδώ τώρα. Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Άντωνη Γουίλεν που είναι επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου της ε, Επιτρόπου κυρίας Νέλης Κρούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα. Καταρχάς να ε, ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κρός, ε, της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής, ε, διότι δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και έχει επενδύσει πολλά, αυτό έχει φανεί και τα τελευταία χρόνια εξάλλου. Έχει επενδύσει ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού της κεφαλαίου. Ο λόγος για τον οποίο ε, δεν είναι εδώ σήμερα είναι γιατί πηγαίνει στο Μπακού αυτή τη στιγμή ε, όπου θα θέσει ρητά τους όρους ε, και τα πρότυπα για την ελευθερία του τύπου, όχι μόνο με το, στον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν τον ίδιο, αλλά και με ε, δημοσιογράφους και ε, όσους ασχολούνται ενεργά με το θέμα της ελευθερίας ε, του τύπου, διότι το Αζερβαϊτζάν ε, πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια πολύ ταραγμένη χώρα όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Τους δημοσιογράφους τους κατασκοπεύουν, τους φυλακίζουν, τους επιτίθενται και η Αντιπρόεδρος Κρούς θα καταδικάσει με πολύ αυστηρούς όρους αυτούς τους περιορισμούς και θα ζητήσει να ληφθούν μέτρα διαφάνειας. Όμως το πρόβλημα δεν είναι θέμα ε, εξοκοινωτικό πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στην, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να δούμε και τις εκθέσεις, ε, τις οποίες ανέφερε και η κυρία Γαβριλίδη. Οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χαίρουν ε, ένα μεγάλο, σε ένα μεγάλο βαθμό την ελευθερία του τύπου. Όμως, σε μια ένωση 27 χωρών υπάρχουν ακόμα προκλήσεις για να έχουμε πραγματικά ένα ανοιχτό και πλουραλιστικό περιβάλλον. Θέματα όπως η συγκέντρωση του τύπου, η ποικιλομορφία του, ο περιορισμός στα ΜΜΕ online και offline, ο έλεγχος, η πίεση, η παρέμβαση από τα κράτη ή πολλές φορές και η, ο απουσία ελέγχου είναι προβλήματα που μας δημιουργούν πίεση. Και η Κομισιό θα παρακολουθήσει ακριβώς τι ε, γίνεται ε, μας ανησυχούν ε, ας πούμε ε, όσα έχουν γίνει ε, στην Ουγγαρία, παρακολουθούμε την κατάσταση εκεί, η Αντιπρόεδρος Κρούς είχε πάει στο Κοινοβούλιο, επίσης και στην Σόφια πήγε πρόσφατα, όπου ήρθε σε επαφή και με τους δημοσιογράφους για την κατάσταση στα βουλγαρικά μέσα μαζικής ανημέρωσης. Επίσης έκανε και μια συζήτηση και με τον Πρωθυπουργό για τις δηλώσεις που έκανε όσον αφορά την διαφορά και επίσης το Κοινοβούλιο πέρυσι ε, εξέφρασε μάλλον ε, τις, ανησυχί, τις ανησυχίες του για τα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία και την Εστονία. Δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχουν σημαντικές ε, και περίβλεπτες αν θέλετε ε, υποθέσεις που παρουσιάζουν την κατάσταση που επικρατεί και στην τομέα της ελευθερίας και στον τομέα του πλουραλισμού του τύπου. Και η Αντιπρόεδρος επανέρχεται με μεγάλη χαρά στο Κοινοβούλιο, αλλά κάθε φορά όμως παρουσιάζει και μια νέα σοβαρή περίπτωση που εμφανίζεται στα κράτη-μέλη και θέλει να ε, συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις στα κράτη-μέλη που κινδυνεύουν να παραβιάσουν κοινέ αξίες, όμως καλό θα είναι να προβλέψουμε την κατάσταση. Και το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκείς αρμοδιότητες για να υπερασπίσει την ελευθερία του τύπου στα κράτη-μέλη. Και αυτή είναι μια ερώτηση που έθεσε και η Αντιπρόεδρος Κρούς διότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από πλευράς της Κομισιό ε, γιατί θεωρούμε ότι έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις ε, καταστάσεις που προκύπτουν στα κράτη-μέλη. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις προσδοκίες και σε αυτά που μπορεί ουσιαστικά και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει η Κομισιό να κάνει και ε, καλωσορίζουμε την πρόσκληση ε, από πλευράς του Κοινοβουλίου να παραστούμε σε αυτή τη συζήτηση, την οποία να παρακολουθούμε πολύ κοντά. Όμως, οποιαδήποτε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτήσει και κάποιες νομικές αρμοδιότητες που θα χρησιμοποιούν, που θα στηρίζονται σε μια επαρκή νομική βάση. Εμείς ε, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό όσον αφορά δηλαδή τις αρμοδιότητες και θα πρέπει να δούμε πώς θα περιοριστεί αυτό το κενό ανάμεσα στις προσδοκίες που υπάρχουν και στις ουσιαστικές αρμοδιότητες. Ξέρω ότι στο σχέδιο έκθεσης κυρίας Βέμπερ αναφέρεται αυτό το θέμα των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν στον τομέα του πλουραλισμού και της ελευθερίας του τύπου. Εμείς ε, ζητήσαμε και από το κέντρο για, τα, για τον πλουραλισμό των, του τύπου και της, την ελευθερία του τύπου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας να αναλύσει τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και υπάρχει και η ομάδα υψηλού επίπεδου την, ε, της οποίας ε, προεδρεύει ο καθηγητής ε, Βάικε Φράιμπεργα, που είναι ο πρώην πρόεδρος της Λετωνίας, ε, και αυτός θα... Και αυτή η κυρία μάλλον ε, θα εξετάσει και το όλο θέμα και θα υποβάλει προτάσεις. Επίσης δεν μπορούμε όταν συζητάμε τα θέματα αυτά να αγνοήσουμε και την, την οικονομική σημασία αυτού του τομέα και έχουν, έχει αλλάξει η οικονομική σημασία. Η Αντιπρόεδρος κυρία Κρούσου δημιούργησε αυτό το φόρουμ για το μέλλον των ΜΜΕ που εξετάζει τις προκλήσεις και τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν και έχει σαν σκοπό να υποβάλει σαφείς συστάσεις για το μέλλον έτσι ώστε δηλαδή να εξασφαλίσουμε την ποικιλομορφία, την ελευθερία και τον πλουραλισμό ε, και να ε, διασφαλίσουμε και την επιβίωση των ΜΜΕ βέβαια από την άλλη πλευρά. Άρα χρειάζεται να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις αξίες, τις αρχές. Δηλαδή, Χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ελευθερία και τον πληραλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο πρέπει να το κάνει αυτό και ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει όντω να υπάρξει μια μεγαλύτερη συσσωρευμένη, αν θέλετε, ε, αθρηστική νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει μέρος σε αυτή τη συζήτηση και όταν ολοκληρωθεί η έκθεση, περιμένουμε με ανυπομονησία να απαντήσουμε σε αυτήν. Ευχαριστώ. Τώρα... Από ό,τι καταλαβαίνω, είχαμε προβλέψει μια παρουσίαση βίντεο τώρα, ε, αλλά θα αντικατασταθεί από την κυρία Νικόλα Φρανκ. Έτσι, έχει αλλάξει ε, λίγο το πρόγραμμα ε, που είναι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της CBU, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τηλεοπτικών Μέσων του Δημοσίου Τομέα από 74 μέλη αποτελείται, 56 κράτη η δηλαδή είναι όλοι οι δημόσιοι φορείς τηλεόρασης στα κράτη-μέλη και αλλού. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Η ελευθεροτυπία που είναι το σημερινό μας θέμα συνδέεται με την πολυφωνία του τύπου στενά. Η ελευθεροτυπία σημαίνει ότι θα υπάρχει εκδοτική ανεξαρτησία, προστασία των δημοσιογράφων και απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια ποικιλία πηγών ενημέρωση. Η πολυφωνία του τύπου σημαίνει ότι οι πολίτε έχουν ευρέως φάσματο πληροφόρηση, γνώμε και απόψεις και δεν ε, θέλει κανεί να επηρεάσει τα πολιτικά ε, ζητήματα από τους φορείς του τύπου. Και αυτά είναι σημαντικά και θεμελιώδη για μια δημοκρατία. Ε, έχουμε ε, πολλές μορφές τύπου, γραπτός τύπος, ηλεκτρονικός τύπος, διαδικτυακός τύπος, ε, με μια μεγάλη πολυφωνία οποιαδήποτε απειλή στην ανεξαρτησία και στη διάθεση αυτών των μέσων, των media, είτε μετά από κυβερνητική παρέμβαση, εκφοβισμό δημοσιογράφων, αδιαφάνεια στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας ή εσκεμμένη απόπειρα ε, μπλοκαρισμού στην πρόσβαση είναι παραβίαση και τραυματισμός της ελευθερίας και της πολυφωνίας του τύπου. Αλλά κάθε μέσο, ε, κάθε media και κάθε χώρα αντιμετωπίζει αυτέ τις προκλήσει και αυτέ τι απειλέ. Ε, συχνά. Ε, τι γίνεται ε, λοιπόν εκεί με τη δημόσια τηλεόραση και ποιος είναι ο ρόλος της. Έχει σημαντικό και κρίσιμο ρόλο για την πολυφωνία του τύπου και αυτό ορίζεται στο πρωτόκολλο της Συνθήκης της Ένωσης για το σύστημα των δημοσίων μέσων ενημέρωσης στα κράτη-μέλη. Είναι το λεγόμενο πρωτόκολλο του Άμστερνταμ γιατί ήταν στη συνθήκη του Άμστερνταμ και τονίζει ότι η ε, δημόσια τηλεόραση συνδέεται στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας και θα πρέπει ε, να γίνεται σεβαστή, καθώς επίσης και η πολυφωνία του τύπου. Η πολυφωνία του τύπου και η ελευθεροτυπία είναι στην καρδιά της δημόσιας τηλεόρασης. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση EBU ε, ενέκρινε μία δήλωση για τις βασικές αρχές και αξίες. Τι ορίζει αυτή η δήλωση, ότι θέλουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο ε, και να εγγυηθούμε την ελευθερία της έκφρασης και να ε, μοιραζόμαστε απόψεις πλουραλιστικές με πολυφωνία. Τονίζει επίσης ε, την ανάγκη να δημιουργηθεί μια κοινή γνώμη, μια δημόσια σφαίρα όπου να γίνονται συζητήσεις. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται το σωστό κλίμα για να ανθίσει αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστή ε, με ε, πολύ σχολαστικό τρόπο η ανεξαρτησία των ε, δημοσίων φορέων ε, ραδιοτηλεόρασης και να έχουν ε, προβλεψιμότητα και ε, στη χρηματοδότησή τους και εγγύηση για τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανεξαρτησία. Η χρηματοδότηση της δημόσιας τηλεόρασης πώς θα γίνει όμως όταν είναι τα οικονομικά δύσκολα. Δυστυχώς κάποιες κυβερνήσεις μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση και να πιέσουν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να αυξήσουν και την επιρροή τους για την εκδοτική γραμμή που θα τηρούν. Αυτό κανονικά δεν πρέπει να συμβαίνει σε μια δημοκρατία κοινωνία. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου του 2010 με τίτλο «Δημόσια τηλεόραση ε, στη ψηφιακή εποχή» ε, τονίζει τις και επαναβεβαιώνει τις ε, απαραίτητες αρχές. Η δημόσια τηλεόραση χρειάζεται δημόσια χρηματοδότηση, επαρκή συμμετοχή σε νέες πλατφόρμες, νέα τεχνολογία και ένα σταθερό περιβάλλον, ρυθμιστικό και κανονιστικό και προβλέψιμο για να υπάρχει υψηλό επίπεδο ειδήσεογραφικό και πολιτιστικό. Επίσης θα πρέπει να διατηρηθεί και η δημόσια ασφαίρα αυτή στην κοινή γνώμη για να είναι ένα σημείο αναφοράς όπου τα blog και τα κοινωνικά δίκτυα ε, δίνουν ε, πολλές ε, πηγές ενημέρωσης. Αλλά δεν μπορεί η κοινωνία να βασίζεται μόνο σε blog, σε Twitter και στη δημοσιογραφία των πολιτών. Ε, χρειάζονται ε, και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ε, που συνεργάζονται με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ακριβώς για να παραμένουν σε επαφή όμως και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι με τα ενδιαφέροντα των πολιτών αυτό ε, το θέμα των social media μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικουρικό αλλά όχι ως υποκατάστατο της πραγματικής δημοσιογραφίας και θα πρέπει να ισχύουν και κανόνες εκεί γιατί η αμεροληψία ε, στη δημοσιογραφία και η ερευνητική δημοσιογραφία είναι στο κέντρο της δημόσιας τηλεόρασης. Τα δημόσια μέσα παίζουν ένα ρόλο για την κοινωνία και αυτό θα φαίνεται και πρέπει να φαίνεται από την πολιτική και από την νομοθεσία των κρατών. Οι θεσμικές εγγυήσεις επιτρέπουν ε, στα δημόσια μέσα να έχουν έχουν πρόγραμμα υψηλής ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ε, προσδοκίες ε, του κοινού με πολυφωνία, με πλουραλισμό, με πολυμορφία που να απευθύνεται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ε, επίσης να λογοδοτεί στο κοινό. Γιατί τελικά ε, η δημόσια τηλεόραση ανήκει στους πολίτες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της CBU ε, δίνει τη δυνατότητα και τονίζει το δημοκρατικό ρόλο ε, των δημοσίων μέσων ενημέρωσης στις χώρες διεύρυνσης και τονίζει και τη σημασία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης για την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται με αυτό το μνημόνιο ε, κατανόησης ε, να τηρήσει το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ και τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γνωρίζετε ότι ήταν πολύ ενεργό σε αυτή την προσπάθεια για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και ορίζει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία, για τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης κτλ. Η EBU επίσης έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις ε, χώρες διεύρυνσης και τους ομολόγους σε όλα τα επίπεδα και στην κατάρτιση και στη στήριξη οικονομική και τεχνική και γενικότερα. Τέτοια μέσα μπορούν να αναπτυχθούν για να τονωθεί και να υποστηριχθεί και στην Ένωση ε, το θέμα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Έχουμε όλο και περισσότερη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης με την τεχνολογία, με την παγκοσμιοποίηση και η κατάσταση γίνεται ε, όλο και πιο περίπλοκη και καμιά φορά όλο και πιο αδιαφανής. Ανταγωνισμό ισχύει ε, εμπορικό και αυτό μειώνει σε κάποιο βαθμό τη συγκέντρωση, αλλά έχουμε συγχωνεύσεις, εξαγορές και έτσι δεν διασφαλίζεται η πολυφωνία του τύπου. Μεγαλύτερη διαφάνεια λοιπόν στα ιδιοκτησιακά των μέσων ενημέρωσης για τους πολίτες ε, θα βελτιώσει ε, τη ε, δυνατότητα της κρίσης για το κατά πόσο υπάρχει πολυφωνία. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πολυφωνία και ο του Ε, για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον ψηφιακό είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες και στο περιεχόμενο ε, μια σωστή πολιτική για το ραδιοτηλεοπτικό φάσμα και με ε, ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο. Ε, τέλος, ε, συνοψίζω. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης παίζουν ένα ρόλο καθοριστικό και σημαντικό για την εγγύηση της ε, ελευθερίας της γνώμης, για την εξασφάλιση της πολυφωνίας και του να ακούγονται όλες οι απόψεις, για να δημιουργείται μια δημόσια σφαίρα, μια δημόσια κοινή γνώμη που να δημιουργούνται εκεί απόψεις και ιδέες, αλλά χρειάζεται η σωστή ε, νομοθεσία, ε, το πλαίσιο, ε, δεδομένη χρηματοδότηση, εξασφαλισμένη και προβλέψιμη για να υπάρχει εκδοτική ανεξαρτησία. Η πολιτική υποστήριξη σε κοινοτικό επίπεδο τι σημαίνει. Αυτό ορίζεται στο μνημόνιο κατανόησης και είναι πρόσδεκτο. Σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχει ένα μέσο για μάλλον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέσο για μεγαλύτερη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και να γίνονται έλεγχοι ε, στη μελέτη σκοπιμότητας για νέα νομοθεσία όταν αυτό χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρος. Ακούσαμε και τους τρεις και τώρα αρχίζει η συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής. Σκεφτείτε και το χρόνο, έτσι. Προτείνω λοιπόν κάθε μέλος που θα λάβει το λόγο να έχει ένα δίλεπτο και μετά να απαντήσουν τα μέλη του πάνελ για να μπορέσουμε να περάσουμε και στον επόμενο γύρο. Η κυρία Αντίτσεβιτς. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you, Honorable. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η δημόσια εμπιστοσύνη στο μέσο, στα μέσα μαζικής ενημέρωση ε, δεν είναι και τόσο μεγάλη και οι λόγοι είναι πολλοί. Ο βασικός λόγος είναι ε, υψηλός βαθμός ε, ανακριβίων, αυτό εντυπωσιακές ειδήσει χωρίς να έχουν κανένα, καμία ουσία και τεράστια περιθώρια κέρδους. Υπάρχει μία τάση ο τύπος να ε, προβάλλει ιστορίες ε, έτσι εντυπωσιασμού, ε, σκάνδαλα σεξ, απαγωγές, όχι ουσιαστικές ειδήσει δηλαδή. Και ε, ενώ ο τύπος απασχολείται με την κάλυψη τέτοιου είδους ε, εντυπωσιαστικών, αν θέλετε, ε, θεμάτων, οι πραγματικές ειδήσει δεν καλύπτονται. Επομένως, η αξιοπιστία του τύπου πέφτει και οι, οι, ειδήσει που αφορούν τις κυβερνήσεις ε, περιορίζονται, ενώ οι ειδήσει ε, που αφορούν τους διάσημους ε, πολλαπλασιάζονται. Επομένως, Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι πρέπει να μαθαίνουμε αντίθετα τι συμβαίνει, τι κάνουν οι κυβερνήσεις, διότι οι κυβερνήσεις ε, ε, ρυθμίζουν τη ζωή μας, μπορούν να μας οδηγήσουν σε πόλεμο. Άρα πρέπει να στρέψουν τα μέσα μαζική ενημέρωση την προσοχή τους σε αυτές τις ειδήσει. Ο τύπος είναι υποχρεωμένος να γράφει την αλήθεια. Τίποτε άλλο εκτό από την αλήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μωράης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταρχάς, η, ευκαιρία που μας δίδεται να έχουμε την έκθεση της Ρενάτα είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι η έκθεση αυτή δίνει και κάποια εργαλεία στην Κομισιό για να αντιμετωπίσει καταστάσεις και αυτές που είχαμε στην Ουγγαρία. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο έθιξε ο Άντωνι Βίλεν, που είναι το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες και στις αρμοδιότητες. Και αυτό το χάσμα ε, είναι η αναπόφευκτη συζήτηση, αν θέλετε, που θα γίνει με βάση αυτά τα θέματα, διότι υπάρχει το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι ζωτική σημασίας και ε, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την, ε, τον πλουραλισμό και την ε, ποικιλία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, υπάρχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία συζητάμε εμεί εδώ σε αυτή τη δική μας επιτροπή και τα θέματα ανταγωνισμού, πολιτικής ανταγωνισμού και πλουραλισμού. Και Εκεί η Κομισιό έχει εργαλεία στο πλωστάσιό της. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα μένα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία για το πώς η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει ε, ορισμένα θέματα, σαν και αυτά που έχουν ε, προκύψει στη δική μου χώρα, παραδείγματο χάρη, διότι εκεί υπήρχε μια μαζική απουσία αυτορύθμισης οι πολίτες ζητάνε όμως μια λύση, απαιτούν μια λύση και αυτή η λύση μπορεί να είναι μια υποχρεωτική νομοθεσία. Και αυτό συμβαίνει στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Κάποιοι πολίτες όμως τρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι αναγκαστικά για την ε, υιοθέτηση υποχρεωτικών λύσεων, αλλά για πράγματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει. Τώρα βέβαια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και μια νομική βάση και δεν ε, είναι ο χρόνο βέβαια για ομιλίε αυτή τη στιγμή, είναι ο χρόνο για ερωτήσει. Γι' αυτό απευθύνω μια ερώτηση στην Κομισιόν. Τι θα γίνει με αυτή την έκθεση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια νομική βάση για να δούμε πώ θα χρησιμοποιήσουμε την πολιτική ανταγωνισμού και να ψάξουμε να βρούμε ένα σωστό νομικό πλαίσιο για το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική ανταγωνισμού για να ε, λύσουμε το θέμα της ε, ε, συγκέντρωση του τύπου. Δηλαδή τι θα κάνουμε για την... ε, συγκέντρωση του τύπου και για τα μονοπόλια του τύπου, τα οποία πλήττουν ε, την ποιότητα των ε, ειδήσεων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, πλήττει αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση προτύπων είναι πολύ σημαντικό θέμα, βέβαια, και δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που θα προκύψουν από την έκθεση αυτή. Όμως πρέπει να υπάρξει με βάση αυτή την έκθεση ένας μηχανισμός ελέγχου. Και θα ήθελα να ακούσω και από την Ρενάτε ποια είναι τα άλλα στοιχεία της έκθεσης ε, τα οποία πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Με Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Γαλλία φέτος ποινικοποίησε ποινικοποίησε ε, επιθέσεις ε, κατά των δημοσιογράφων και επίσης τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ορισμένες άλλες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ποινικοποίησει διαστρέβλωση ιστορικών γεγονότων και πιστεύω ότι τέτοια γεγονότα, τέτοιες αποφάσεις ποινικοποίηση δεν συνάδουν με την ελευθερία του τύπου, των μέσων ενημέρωσης, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν βίες αντιδράσεις. Ο περιορισμός ε, των, της έκφρασης δεν είναι αποδεκτός. Κάθε προσπάθεια περιορισμού ε, πρέπει πρόσφατα ε, ε, να δούμε πόσες χώρες προσπαθούν να περιορίσουν την ελευθερία του διαδικτύου και να κλείσουν ε, υπηρεσίες προσφοράς υπηρεσιών του διαδικτύου σε τρίτες χώρες, σε άλλες χώρες. Πολλές φορές ε, οι πράξεις αυτές ε, γίνονται χωρίς αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, διότι δεν υπάρχουν οι νόμοι δίωξης. Ο περιορισμός ε, κατά των μέσων έκφρασης αυτομάτως δημιουργεί και ένα περιορισμό ανάγνωσης και ακρόασης και πρόσβασης. Στη Γερμανία φέτος έγινε μία συζήτηση για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 Ναι. τον, την απαγόρευση ενός πολιτικού κόμματος και άκουσα τις απόψεις όλων των πολιτικών κομμάτων εκτός βεβαίως από το κόμμα αυτό το οποίο η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει. Ε, ακόμα πιο προβληματική είναι η νόμη κατά της ελευθεροτυπίας ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ε, δεν υπάρχει καμία ε, άμυνα αυτού, αυτής της απόφασης, καμία δικαιολογία. Ευχαριστώ. Ε, ε. Κυρία Γκιόνς, ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε μια σειρά διλημάτων εδώ και από τους συζητητές ακούσαμε και από τους ομιλητές μας. πιστεύω όμως ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία για να πούμε ότι είναι καλύτερη η Ευρώπη από άλλα μέρη του κόσμου ως προς την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας και να κάνουμε και μαθήματα σε άλλες χώρες και να δίνουμε συμβουλές, τότε θα πρέπει κάπως να τηρούμε και τις προσδοκίες ε, που υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ρηφθεί υπόψη ε, βεβαίως και τις αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Το κατανοώ αυτό και πολύ σημαντικό να σεβόμεθα τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των θεσμικών οργάνων. Ε, να μην παραβιάζουμε τα όρια αυτά. Αλλά ε, ελπίζω ειλικρινά να έχουμε και περισσότερες ευκαιρίες με τη συνθήκη της Λισαβόνας να ε, υπερβούμε τους ε, πρόσφατους κανονισμούς. Και επίσης βεβαίως δεν χρειάζεται υπερβολική ρύθμιση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφορετικότητα, πολυμορφία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα αξιοπιστίας εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδοκιών των πολιτών μας. Και αυτά είναι πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο. Όσο μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Περιμένω ε, την έκθεση που ανέφερε ο κ. Γουίλαν της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου. Πρόσφατα το συζητήσαμε, αρχίσαμε να συζητούμε αυτά τα θεμάτα και να δούμε τι θα υποβάλει στην κυρία Κρού, στην επίτροπο αυτή η ομάδα. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε αρκετό θάρρος για να πούμε κάτι και στην έκθεση αυτή και αλλού και να υπάρχει κάπου ουσία στις συστάσεις ε, της ομάδας υψηλού επίπεδου. Και να ε, ξεπεράσουμε τις πρόσφατους κανονισμούς, την πρόσφατη ρύθμιση. Η κατάσταση είναι όλο και πιο επικίνδυνη. Δεν αρκεί να κάνει τη δουλειά του το Συμβούλιο της Ευρώπης ή ο ΑΣΕ. Ε, θα πρέπει να βγει κάτι δεσμευτικό από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και υπάρχει ιδιαίτερη εδώ ευθύνη από όλε τι πλευρέ των ε, κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα προηγουμένως, ε, έπρεπε να είμαι σε άλλη επιτροπή. Ε, μου είπαν διάφορα υπάλληλοι και οι συμβουλοί που υπόθηκαν. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που ε, είπαν και οι προλύσαντες και η κυρία Γκιόνς τώρα μόλις. Πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου η Ένωση στο εσωτερικό της, στα κράτη-μέλη της. Αυτό είναι σημαντικό και προς το εξωτερικό. Εγώ πηγαίνω στα Δυτικά Βαλκάνια και μιλάω εκεί για ανεξαρτησία τύπου, για τους δημοσιογράφους που θα πρέπει να έχουν ελευθερία και να αντιμετωπίζουν και κρίσιμα ζητήματα. Κάθε φορά που τα λέμε αυτά ακούμε... Ναι και στο εσωτερικό της Ένωσης τι γίνεται, ε, είναι τα πράγματα όσα οφειλάν, ε, τι επικρατεί εκεί. Και θέλω να υποστηρίξω αυτούς που ζητούν υψηλό επίπεδο όχι μόνο ελέγχου και παρακολούθησης, αλλά πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κάποια στοιχειώδη ε, πρότυπα ελευθερίας του τύπου. Και θέλω να ακούσω ε, από σας μια απάντηση. Βέβαια αυτό θα μπει και στην έκθεση της Ρενάτε Βέμπερ, αλλά τι μπορούμε να σκεφτούμε για να το ρυθμίσουμε. Μπορούμε να έχουμε δεσμευτικά πρότυπα. Και αυτό τι σημαίνει μετά για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και αν υπάρξει μια παραβίαση αυτών των κανόνων και των προτύπων. Θα ακολουθήσουν και κυρώσεις. Ξέρω ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό, αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε εκείνοι που θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα που ήθελα να σας υποβάλω και ακριβώς ότι θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και στους πολίτες μας και στον εαυτό μας αλλά και στους πολίτες τρίτων χώρων. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρινέσκο. Ε, ε, ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε όταν μιλάμε για την ελευθερία του τύπου είναι η παρέμβαση των κυβερνήσεων ή παρέμβαση κρατική. Αυτή τη στιγμή όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι τα μέσα αυτά ελέγχονται ε, με βάση τις πολιτικές ε, προτιμήσεις των ιδιοκτητών τους. Τι προτίθεστε να κάνετε σε αυτό το θέμα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η έκθεση αναφέρεται σε μια πιθανή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω της θέσπισης ε, σχετικής νομοθεσίας. Τι έχετε κατά νου. όταν αναφέρεστε σε αυτή την πιθανή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και κάτι τελευταίο. Είναι αλήθεια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι ελεύθερα. Από την άλλη πλευρά όμως και οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι ελεύθεροι μεν, αλλά να σέβονται έναν κώδικα διοντολογίας δηλαδή ελεύθεροι από πιέσεις ε, που θα προέρχονται από τους ιδιοκτήτες των μέσων μεζικής μέρους, από τον χρηματισμό, από την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να σέβονται όμως, να αυτοδεσμεύονται από ένα κώδικα διοντολογίας. Ποια είναι τα σχόλιά σας. Κύριε Μάκιντάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμμετέσχουν μέχρι τώρα και παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Βίλαν. Ιδίω εκεί που ανέφερε τις απρόσμενες επιπτώσεις, αναπάντεχες επιπτώσεις και ότι πολεμούμε κατά του, του νόμου των απροσδόκητων επιπτώσεων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτόν τον, την πτυχή. Πρέπει καταρχάς να εξετάσουμε που πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν ήδη συμφωνίες πλαίσιο που έχουν υπογραφεί, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με την υλοποίησή τους και πού μπορούν να βελτιωθούν. Δεύτερον, πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητες και πού έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς, το οποίο έχει τονιστεί ήδη προπηγούμενους ομιλητές. Όσον αφορά στο ερώτημα της ενιαίας αγοράς και αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομοθεσία των κρατών μελών αποτελεί ένα πρόσκομα ε, στους κανόνες του σεμιτού ανταγωνισμού και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Προέρχομαι από το Ενωμένο Βασίλειο και γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και είναι σημαντικό να δούμε την ισορροπία μεταξύ ελευθεροτυπίας και ευθύνης των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία. Επίσης, μαζί με τη Ρενάτε Βέμπερ, ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την Ουγγαρία και παρόλο που η Ουγγαρία αναφέρεται σχετικά με την ελευθεροτυπία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ε, πρέπει να δούμε ότι η έκθεση αυτή θα καλύψει όλο το φάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή δεν στοχεύει μόνο στην Ουγγαρία. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε επίσης πιο πολύ σημασία στην ευθύνη των μέσων ενημέρωσης. Ο πρόεδρος, επανέρχομαι τώρα στους, στα μέλη του πάνελ, η κυρία Γαβριλίδου. Ε, θα ήθελα να πάρει το λόγο πρώτη, πρώτη να απαντήσει. Ας ε, ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία uh, There is a dilemma here. με τον κύριο Μπρόνς. Ε, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, πρέπει να ρυθμίσουμε αλλά όχι να υπερρυθμίσουμε, να ρυθμίσουμε δηλαδή υπερβολικά. Πρέπει να κρατήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο απλό, ε, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία να προσέξουμε την ε, απλούστευση. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργούμε περιπλοκότητες, αλλά πολύ πιο, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργούμε περιπλοκότητες, πολύ πιο δύσκολο να κρατάμε τα πράγματα απλά. Βεβαίως και εγώ ενδιαφέρομαι για την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ε, η ελευθερία ε, των μέσων ενημέρωση σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές του νομίσματος λειτουργούν. Αλλιώς δεν γίνεται. Και πολλές φορές ε, αυτά που ακούς επικεντρώνονται στις, ε, στο κράτος, στις κυβερνήσεις, ε, στους δημοσιογράφους και βεβαίως ο δημοσιογραφικός κόσμος εξαρτάται από πλευράς μισθού, από τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης αλλά δεν είναι αυτό το μόνο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης και ίσως αυτό το πρόβλημα διονγκώνεται υπερβολικά. Ε, οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι, φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, κλείνουν σταθμοί, κλείνουν μέσα ενημέρωσης, οπότε είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν ακριβώς αυτά που ζητάνε τα αφεντικά τους, οι ιδιοκτήτες αν θέλετε. Ε, βεβαίως πρέπει να τους προστατεύσουμε λοιπόν με ένα πλαίσιο το οποίο είναι απλό, εφαρμόσιμο, εύκολο να εφαρμοστεί και εύκολο να το εποπτεύσουμε. Ο κύριος Βίλαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάρα πολλά ε, θέματα τέθηκαν και θα ήθελα να απαντήσω σύντομα. Καταρχάς ο κύριος Μωράες ε, έσυξε ένα σημαντικό θέμα διότι είπε ότι πολλά ξεχωριστά θέματα έχουν δεσμευτεί υπό την ομπρέλα, υπό το γενικό θέμα του πλερισμού. Ε, και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε τα μέσα έτσι ώστε το κράτος να κρατιέται σε απόσταση αλλά ε, επίσης να δίνεται η δυνατό, διότι βλέπουμε ε, αυτή τη στιγμή να υπάρχουν παρεμβάσεις και μάλιστα ισχυρές σε ορισμένα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει ακριβώς να ξέρουμε τι θέλουμε, τι επιδιώκουμε. Στον πλουρισμό, στη διαφάνεια, στην ανεξαρτησία όσον αφορά δηλαδή τι δημόσιε ρυθμιστικέ αρχέ Και όταν λέμε ανεξαρτησία, τι ακριβώς στοχεύουμε, ε, όταν υπάρχουν φαινόμενα συγκέντρωσης ε, της τέταρτης εξουσίας. Όσον αφορά τώρα τα ερωτήματα αυτά για τις αρμοδιότητες δεν είναι ασαφείς. Ε, θέλουμε να ξέρουμε, έχουμε την αρμοδιότητα να επιτελέσουμε το α, β ή γ. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, εξετάζουμε και το θέμα των αρμοδιοτήτων παράλληλα με το θέμα των επιδιώξεων. Στην Κομισιόν θεωρούμε ότι δεν έχουμε πλήρη ελευθερία δράσης επειδή κάτι αναφέρεται στον ε, χάρτη των δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο λειτουργικό για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ουσιαστικές διατάξεις. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, ο υπάρχον, ε, υπάρχουσα νομοθεσία βεβαίως είναι απόλυτα σχετική, αλλά όταν ε, προσάπτονται κατηγορίες ε, αποτυχίας της αυτορύθμισης και πολύ σωστά θα πρέπει να εξετάζουμε και το θέμα της ιδιωτικότητας ε, των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Άρα χρειάζεται να προσέξουμε το, το υπάρχον πλαίσιο προστασίας και να δούμε εάν εφαρμόζονται σωστά οι υπάρχουσες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επιλύσουν ένα μέρος των προβλημάτων. Όσον αφορά ε, αυτά που είπε η κυρία Λούνατσεκ για την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων για την εποπτεία ε, και, την, ε, και τον έλεγχο και αυτό πάλι βεβαίως επισέρχεται στον τομέα των αρμοδιοτήτων αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί βεβαίω η συζήτηση. Θέλω να δω και την άποψη του συν νομοθέτη, του άλλου νομοθέτη δηλαδή, νομοθετικού σώματος. Ε, πρέπει να βρούμε λειτουργικούς τρόπους για να εφαρμοστούν πρακτικά οι διατάξεις και όχι ακαδημαϊκά. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα τα, τα πολλά από τα απαραίτητα λειτουργικά εργαλεία στα χέρια μας. Επίσης, απαντώντας στην παρατήρηση της κυρίας Αντίτσεβιτς, όταν ε, εξετάζουμε διάφορα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης και το υλικό που χρησιμοποιούν, είναι δύσκολο όταν μιλάμε για ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να πούμε ότι ένας μία μορφή είναι νόμιμη και άλλη δεν είναι. Από πλευράς τώρα όμως κοινού πρέπει να μελετήσουμε τις οικονομικές συνθήκες που θα επιτρέπουν ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης να λειτουργεί αποτελεσματικά με τις παρούσες συνθήκες. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρονται αυτά τα θέματα στην έκθεση για το μέλλον των μέσων ενημέρωσης. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Η κυρία Φρανκ, ευχαριστώ. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε και αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένας βαθμός απογοήτευσης ε, μεταξύ των μελών μας. Εγώ ανέφερα το μνημόνιο e το μνημόνιο κατανόηση. και ελπίζω τα μέλη μας να ιδίω στις, στις νέες χώρες μετά την διεύρυνση να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την και, να αγκαλιάσουν αυτή τη δέσμευση. Είναι μια πολύ βαριά απέτηση αυτή που έχουμε από την Κομισιόν, αλλά αυτή η δραστηριότητα, αυτή η ενεργό συμμετοχή της Κομισιόν και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων σταματάει εκεί όπου δεν υπάρχουν αρμοδιότητες. Ε, ε, το κανονιστικό πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης είναι, ε, είναι στα χέρια των εθνικών αρχών και γι' αυτό υπάρχει ακριβώς αυτός ο βαθμός απογοήτευσης όλοι λέμε ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει νομική βάση για οποιαδήποτε παρέμβαση και πρέπει αυτό το πλαίσιο των κανόνων και των ρυθμίσεων ε, να είναι χρήσιμο ε, έτσι ώστε να βοηθάει και να ενισχύει τον πλουραλισμό ε, και οι μελλοντικές ρυθμίσεις, αυτές που είναι εν και οι μελέτες επιπτώσεων πρέπει να έχουν αυτό το στόχο πρέπει να εξετάσουμε πιο πολύ βάθος την, ε, τα εποπτικά όργανα, τις εποπτικές αρχές. Ε, αναφέρεται, αναφέρονται ορισμένα σημεία στην έκθεση, αλλά πρέπει να τα εξετάσουμε περαιτέρω. Τη λειτουργία και υλοποίηση του, του έργου των εποπτικών αρχών. Όσον αφορά τώρα ε, τα, τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό διαφάνειας ιδιοκτησίας ε, των ιδιωτικών μέσων για να ξέρουν και οι πολίτες να ξέρει το κοινό ποιος έχει ποια συμφέροντα, εμπορικά συμφέροντα, ιδιωτικά συμφέροντα. Ε, είναι πολύ πιο εύκολο για μας να κρίνουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε εμείς από αυτά τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφερα ότι υιοθετούμε συζητήσαμε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές για τα μέλη μας και όχι μόνο στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε 56 χώρες μέλη και εκτός βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομολογώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ανεξαρτησίας ε, σε πολλές χώρες, ε, όχι μόνο από τις χώρες της διεύρυνσης, αλλά ε, προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, παραδείγματος χάρη θέλουμε να υιοθετήσουν ορισμένες αρχές ε, σύνταξης, συντακτικές αρχές των αρχισυντακτών, δηλαδή τη σύνταξης, και πιστεύουμε ότι είναι μόνο, ε, αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε μόνο σε ένα πολιτικό περιβάλλον που, όπου τα μέσα ενημέρωση λειτουργούν ανεξάρτητα και ελεύθερα. Η εισηγήτρια η κυρία Βέμπερ, πολύ σύντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται, σε, βασι, βασίζεται κυρίως σε, δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά συμφέροντα, αλλά θα έλεγα ότι η βάση της είναι μία βάση αρχών. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να ε, ξεπεράσουμε αυτά τα προσκόμματα τα οποία ε, δεν, είναι, δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το να επιβάλλουμε κυρώσεις, ε, η αλήθεια είναι ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται όταν υπάρχουν παραμβιάσεις, αλλά όταν λέμε κυρώσεις σε εισαγωγικά, εννοώ ότι πρέπει να λάβουμε μία θέση ξεκάθαρη για το πώς ορίζουμε μία συγκεκριμένη κατάσταση σε ένα κράτος μέλος ή σε περισσότερα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εννοώ ότι η έλλειψη νομικών προτύπων, η έλλειψη αρμοδιοτήτων δεν είναι επαρκής δικαιολογία σε περίπτωση παραβιάσεων. Πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι, πρέπει να έχουμε ισχυρή πολιτική βούληση, να πρέπει να να δεσμευτούμε, να αγκαλιάσουμε όλοι ακλόνητα την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Και η ευρωπαϊκή κοινότητα, ε, δεν εννοώ προσωπικά, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, συγγνώμη, δεν εννοώ συγκεκριμένα την Επίτροπο Κρούζ, η οποία έχει δώσει μεγάλες μάχες. Αλλά πολλές φορές η η Κομισιόν τηρεί σιωπή όταν συζητούμε τέτοια σημαντικά θέματα και θα ήθελα να δω μια αλλαγή στάσης στο μέλλον. Αυτό το οποίο μας λείπει είναι μια ισχυρή πολιτική βούληση και το θάρρος ε, να προχωρήσουμε. Στα θέματα της ευθύνης εκεί που είμαι πολύ επιφυλεκτική είναι στο εξής. δεν θέλω να χρησιμοποιηθεί η δικαιολογία των ορμοδιατήτων ως όπλο στα χέρια της κυβέρνησης ε, να εκτελέσει, να επιτελέσει παραβιάσεις και καταχρήσεις εναντίον της ελευθερίας. Ε, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε γνήσιο πλουραλισμό χωρίς διαφάνεια. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική διαφάνεια. Να ξέρουμε ποιος ή ποιοι είναι πίσω από ένα συγκεκριμένο έργο, μια συγκεκριμένη κατάσταση. Όταν θα έχουμε αυτές τις πληροφορίες, τότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των γεγονότων. Αλλά αυτά βέβαια πρέπει να τα συζητήσουμε, διότι είναι ε, και οι κυβερνήσεις υπεύθυνε και έχουν ε, πολλή εξουσία στα χέρια τους. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα και ήταν πολύ επικοδομητικά. Ωραία. Μου λέγουν ότι υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Προετοιμασίες για να δούμε το βίντεο ε, έχουν ολοκληρωθεί και μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Αλλάζει λοιπόν το πάνελ και περνούμε στο επόμενο και θα πρότεινα να αλλάξουμε τη σειρά. Να δούμε πρώτα το βίντεο που είχε ανακοινωθεί. Let's, let's hear as we proceed with the panel. Thank you. Thank you, Mrs. Frank. Okay, yes, yes. Now, now. Λοιπόν, Η κυρία Ντάνια Μιγιάτοβιτς του ΟΑΣΕ θα μας παρουσιάσει το βίντεο. Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για την ελευθεροτυπία. Δυστυχώς ε, κολλείεται και απουσιάζει η κυρία Μιγιάτοβιτς, αλλά μας στέλνει αυτή τη συνεισφορά υπό μορφή βίντεο. Είναι ένα ε, οπτικό-ακουστικό μήνυμα που θα δούμε και καλούμε τους υπολείπους του πάνελ να έρθουν εδώ. Την κυρία Πέγγι Βάλκε από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης. Ο κύριος Μάριος Ντράγκομι που είναι ε, από το Project Mapping Digital Media για την χαρτογράφηση των ψηφιακών μέσων και την κυρία Μάγδα ε, Βάλτερ και θα σου πεις και τον κύριο Ιβαρ Ράσταλ που είναι πρόεδρος των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδοτών Εφημερίδων. Ε, ακούμε λοιπόν την κυρία Ντούνια Μιγιάτοβιτς. Yes? What, what, what about that? Sound problem? Sound problem? Υπάρχει πρόβλημα ήχου. Βλέπουμε την κυρία, αλλά δεν την ακούμε. Can we replay? Ladies and gentlemen, I'm Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω ε, με αυτό το μήνυμα βίντεο στη δημόσια ακρόασή σας για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ελευθεροτυπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Ορίστηκα εκπρόσωπος για την ελευθεροτυπία πριν από μία τριετία. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών είχα αντιμετωπίσει μια σειρά ε, ζητημάτων ε, ελευθεροτυπίας στα 56 κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να δράξουμε την ευκαιρία που έχουμε ενώπιόν μας άμεσα. Να πληρώσουμε τις ε, δεσμεύσεις μας και να δημιουργήσουμε ε, περιβάλλοντα όλα τα κράτη-μέλη που θα δημιουργήσουν, θα θρέψουν και θα βοηθήσουν την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης. Θα ήθελα επίσης να ε, χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να αναρωτηθώ αν όχι τώρα πότε, αν όχι εδώ πού. Διότι αυτή τη φορά, παρόλο που όλες οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει να προστατεύουν και να ενισχύουν την ελευθερία του τύπου, όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής, πολλές χώρες υπολείπονται κατά πολύ των υποχρεώσεων και δεσμεύσεών τους. Πρόσφατα, η κατάσταση έγινε πιο ανησυχητική σε ορισμένες χώρες συμπραγμανωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθεροτυπία, η πολυφωνία του τύπου και η δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση διαβρώνεται χρησιμοποιώ κάθε ευκαιρία που έχω για να αυξήσω την προσοχή και τη φωνή μου σε αυτή την ανησυχητική τάση. Αλλά η δική μου φωνή και μόνο δεν αρκεί για να αλλάξει τίποτα αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να θεωρηθεί η ελευθεροτυπία ως θεμελιώδες δικαίωμα που επιτρέπει στον κόσμο να αλλάζει τις κοινωνίες και να τις κάνει παλόμενες δημοκρατίες ε, και να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τόπος που θα πρέπει να πηγάζουν αυτές οι ιδέες. Και ε, η περιοχή του ΟΑΣΕ θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και ε, καλές πρακτικές για νεοσύστατες αναδυόμενες δημοκρατίες, για να το ακολουθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει μοναδική ευκαιρία να συμπεριλάβει ουσιαστική ελευθεροτυπία ως κριτήριο επιλέξιμο για την ένταξη ε, χωρών υποψηφίων και ενδεχομένως υποψηφίων. Η ηγεσία της Ένωσης δια του παραδείγματος ε, δεν θα είναι μόνο προ όφελο της Ένωσης αλλά ε, θα μπορούμε και στην εξωτερική πολιτική να ζητάμε την ελευθεροτυπία δικαιολογημένα. Ωστόσο στην καθημερινή μου δουλειά βλέπω ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κυβερνήσεις που θεωρούν τα μέσα ενημέρωσης επικίνδυνη πλατφόρμα που θα πρέπει ε, να ελέγχεται και καμιά φορά να φημώνεται. Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουν οι αρχές αυτές ότι αυτή η συμπεριφορά προς τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί παρά να αποδυναμώσει ε, τις δημοκρατικές αρχές που τόσο αγαπούμε και βασίζουμε τις κοινωνίες μας. Πρώτος στόχος είναι, είναι να προλάβω τη βία κατά των ε, δημοσιογράφων, φυσική παρενόχληση, εκφοβισμός, ε, ξυλοδαρμός, ακόμα και ε, φόνοι, δολοφονίες δημοσιογράφων παρατηρούνται. Έχουμε δει και σε διάφορα κράτη-μέλη, Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, ε, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, τέτοια κρούσματα. Οι διώξεις και οι ανακρίσεις προχωρούν αργά και οι δράστες δεν έχουν έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης βλέπουμε και δημοσιογράφους ε, στην Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία να ε, παρενοχλούνται την ώρα που καλύπτουν διαδηλώσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις. Θα πρέπει να ε, προστατεύουν αρχές επιβολής του νόμου τους δημοσιογράφους και να τους επιτρέπουν να κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους. Βλέπω όμως να ασκούνται και πολιτικές πιέσεις στα μέσα ενημέρωσης και κρούω τον του, το κόδωνα του κινδύνου. Και ε, είναι γνωστό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσα να σας πω διάφορες χώρες όπου βλέπω πολιτική πίεση ω σημαντική απειλή για την ελευθερία της έκφρασης. Θα πρέπει όμως εδώ να επικεντρωθούμε στην Ουγγαρία. Από το 2010 ε, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τύπο στην Ουγγαρία έχει αναδιοργανωθεί εκ βάθρων και ανησυχεί βαθύτατα και τη δική μας ε, υπηρεσία και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό όχι για μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνούς θεσμούς να ε, δώσουν ιδιαίτερη σημασία και προσοχή πολύ νωρί και να αρχίσει ένας διάλογος με τις αρχές για να μην προχωρήσει η νομοθεσία που θα επηρεάσει αρνητικά όλες αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, έχει περιοριστεί η πρόσβαση του κόσμου στην ενημέρωση ε, και μεταξύ των 27 κρατών μόνο η Ισπανία, Εστονία, Ιρλανδία, Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αποποινικοποιήσει τη συκοφαντική δυσφήμιση. Σε παλαιότερες δημοκρατίες ε, αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει την ελεύθερη δημοσιογραφία Γενικά όμω αυτά δεν φτάνουν στα δικαστήρια και στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Θα πρέπει όμως να αποποινικοποιηθεί γενικότερα η συγκοφατική της φήμηση γιατί επηρεάζει τον τύπο αρνητικά. Θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε ε, ότι ε, κανένα κράτος δεν εξαιρείται αυτό. Αυτό βλέπουμε από διαδικασίες στην ποινική δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση στην Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία και Πολωνία. Το θέμα δεν είναι μόνο η συγκοφαντική δυσφήμιση. Δεν μπορεί μόνο αυτή να στείλει τους δημοσιογράφους στη φυλακή. Ε, καλωσόρισα την ε, αθώωση του Έλληνα δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη που θεωρήθηκε ότι παραβίασε προσωπικά δεδομένα και ε, η δίκη του δήρυξε μία μέρα. Ε, η απόφαση αναγνωρίζει το βασικό ρόλο που παίζουν τα μέσα ενημέρωσης όταν συζητούν θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Το 2005 το Βέλγιο ε, πέρασε ένα νόμο που εγγυάται ισχυρή προστασία των πηγών που πρέπει να παραμένουν απόρριτες. Θα πρέπει όλες οι αρχές να εξαντλούν ε, όλες ε, τις πηγές πριν ζητήσουν από δημοσιογράφους να αποκαλύπτουν τις δικές τους. Και αυτό να είναι παράδειγμα για άλλους. Στη τσεχική δημοκρατία ένα δικαστήριο επικαλέστηκε απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να μην αποκαλυπθούν πηγές ε, στην αστυνομία. Παρακολουθούμε την νομοθετική διαδικασία και την προπαρασκευή στην Ισπανία για τη διαφάνεια, την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ελπίζω ο νόμος να αντανακλά τις πιο προηγμένες προδιαγραφές και να εγκριθεί σύντομα από την Ισπανική Βουλή. Η ελεύθερη έκφραση και εξασφάλιση της στο διαδίκτυο παρεμένει υψηλά στην ημερήσια διάταξη του γραφείου μου. Βλέπουμε και πάλι ανησυχητικές προσπάθειες των κυβερνήσεων και των αρχών να ή να περιορίσουν. Μα το διαδίκτυο δεν γνωρίζει ε, σύνορα. Ε, δεν θα λυθούν τα προβλήματα ε, από υποτιθέμενα επικίνδυνο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη, περισσότερη εκπαίδευση και γνώση περί τα θέματα του τύπου για να επιτρέπεται η πλήρης ελευθερία της έκφρασης. Και ε, με αυτό το θέμα θα ήθελα να κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δράση του τον Ιούλιο που απέρριψε την άκτα. Η άκτα βασίζεται σε μια κατανοητή επιθυμία ε, να περιορίσει ή να ε, πάυσει και να καταπολεμήσει την παραβίαση του copyright, αλλά δεν είναι η λύση τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να προστατεύονται διαφορετικά. Ε, και πάλι συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, δράσεις και τις ενεργές του. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι επιτυχή συζήτηση, την οποία και θα παρακολουθώ από το διαδίκτυο. Και σας ευχαριστώ και πάλι που με προσκαλέσατε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. I have to say that we have always... Ναι. Πάντα έχουμε πολύ καλές ε, σχέσεις συνεργασίας με την κυρία Ντούνια Μιγιάτοβιτς και την ευχαριστώ. Και περνούμε αμέσως ε, στον επόμενο ομιλητή που είναι ομιλήτρια, είναι καθηγήτρια Πέγγι Βάλκε, καθηγήτρια στο Καθελικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης και ασχολείται με θέματα ελευθεροτυπίας εδώ και καιρό. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βέμπερ. Κυρίες και κύριοι, είναι μια τιμή και ευχαρίστηση για μένα που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και που μπορώ να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου για το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση των ελευθεριών των μέσων μαζική ενημέρωση και του πλουραλισμού στα κράτη-μέλη. Καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία για την υιοθέτηση του ψηφίσματος για τα πρότυπα για την ελευθερία των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα πρώτο βήμα για να ληφθούν ε, πιο συγκεκριμένα μέτρα με βάση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν καθηγήτρια νομικής στα Πανεπιστήμια της Λεβά των Βρυξελών και του Τίλμπουργκ συμμετείχα σε διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ελευθερία του τύπου και τον πλουραλισμό τα προηγούμενα χρόνια. Σαν project leader για την μελέτη για τους δείκτες για τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ ή σαν νομική σύμβουλος ε, για την ε, μελέτη Interreg για τους δείκτες για ανεξαρτησία και αποτελεσματικής λειτουργίας των οπτικοακουστικών μέσων ε, ενημέρωσης. Όπως επίσης συμμετείχαμε και σε μια άλλη ε, συνάντηση, η οποία χαρακτηρίστηκε βέβαια η συνάντηση Hugh Grant, διότι συμμετείχε και εκεί, δεν ήταν όμως μόνο αυτός, ήταν ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ για τον πλουραλισμό στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το ενδιαφέρον μου και ο ρόλος μου σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι καθαρά ακαδημαϊκός. Όταν ε, έχω ξεκινήσει Ε, τις δραστηριότητές μου ε, και στα, στο Φλαμανδικό Κοινοβούλιο και στο Βελγικό Κοινοβούλιο, όμως η οι απόψεις που θα εκφράσω σήμερα είναι καθαρά προσωπικές και θα στηρίζονται στην, ε, στην εμπειρία που έχω. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια ιστορία για να απαντήσουμε στην ερώτηση που με μετέθη. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οδηγία για να εξασφαλίσουμε τον πλουραλισμό. Καταρχάς θεωρώ ότι η ερώτηση είναι σωστή. Έχουμε ε, οδηγίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Όχι. Έχουμε όμως την οδηγία η οποία έγινε κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στα εκτιμώντας λέει ότι έχει σαν στόχο να διασφαλίσει την εσωτερική αγορά μέσα στην οποία τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και στα οποία τα ε, ε, τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα του ατόμου πρέπει να διασφαλίζονται. Ταυτόχρονα έχουμε μία οδηγία, την οποία αναφέρω, που προσπαθεί να δημιουργήσει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις υπηρεσίες του τύπου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και υψηλή προστασία των, των στόχων. Αυτή η οδηγία υπάρχει από το 2089. Είναι η οδηγία τηλεόραση χωρίς σύνορα και μετά με το ονομάστηκε οδηγία οπτικοακουστικών μέσων. Και αυτή η οδηγία καλύπτει όμως κάποιες διατάξεις ε, που έχουν μεταφραστεί με νομοθετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κανονισμούς στα κράτη-μέλη. Επομένως και είναι περιορισμένος, περιορισμένο το πεδίο εφαρμογής της. μιλάμε για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τα media on demand, εκεί περιορίζονται. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διασυνοριακές, κατ' ουσίαν και επομένως υποφέρουν περισσότερο από τις ελλείψεις στις εθνικές νομοθεσίες. Επίσης, αυτές οι υπηρεσίες υπόκεινται σε κρατική νομοθεσία λόγω ακριβώς των συνεπειών που έχουν στο κοινό. Άρα υπάρχει περισσότερη νομοθεσία έτσι ώστε να εναρμονιστούν με βάση την οδηγία για τις ε, υπηρεσίες των οπτικοακουστικών μέσων. Αλλά ποιοι είναι οι λόγοι για να περιορίσουμε αυτούς τους συντονισμένους τομείς ε, σε αυτούς που αναφέρονται τώρα στην οδηγία, δηλαδή η προστασία των ανηλίκων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πολιτιστική ποικιλομορφία, πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, κάλυψη σημαντικών γεγονότων, πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, προστασία του καταναλωτή σε σχέση με τις εμπορικές ανακοινώσεις στην τηλεόραση και το δικαίωμα προς απάντηση. Γιατί αυτή η περιοχή, αυτές, αυτοί οι δεν διευρύνθηκαν ή δεν συμπληρώθηκαν με εναρμονισμένε ε, διατάξει. Παραδείγματο χάρη για την διαφάνεια των, ε, ε, στην ιδιοκτησία των μέσων μαζικής ενημέρωση. συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδιοκτησίας δηλαδή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε, δεν υπήρχε αρμοδιότητα, Εάν ναι, ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί σε αντίθεση η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δίκτυα μάλλον ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, που στηρίζεται επίσης στην, στην λογική της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβάνει κανόνες για την οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία των εθνικών κανονιστικών χωρών. γιατί το πακέτο αυτό ε, επιτρέπει την ε, πρόσβαση στην αγορά για τις ηλεκτρονικές ε, υπηρεσίες. Βέβαια δεν έχουμε πολύ, πολλούς πόρους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό γιατί, διότι θεωρούμε ότι αυτές ε, οι ρήτρε διασφάλισης είναι πιο σημαντικές ε, σε σχέση με τα δίκτυα από, ότι, από το περιεχόμενο. Ε, μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι τηλεφωνικοί λογαριασμοί από την αξιόπιστη και διαφοροποιημένη ενημέρωση. Δεν το πιστεύω αυτό. Επομένως, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την ε, ότι δεν πρόκειται να συμβεί οποιαδήποτε πράξη η οποία θα προωθήσει την δημιουργία ε, κυριάρχου δεσποζουσών θέσεων που θα οδηγήσουν σε περιορισμό του πλουραλισμού και της, στην, ε, ελευθερίας στην ε, τηλεοπτική ενημέρωση και, της, και στην ενημέρωση εν γέννη. Και θα πρέπει ο Ευρωπαίος νομοθέτης ενδεχόμενα να υπερασπίσει την εσωτερική αγορά και να δικαιολογήσει την ανάγκη για τέτοιες ρήτρες διασφάλισης σε σχέση με τα δίκτυα. Μεν, αλλά και κυρίως σε σχέση με το περιεχόμενο. Υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την ιδιοκτησία των ΜΜΕ και όσον αφορά τα κατόφλια, τα όρια δηλαδή, και όσον αφορά τις παραμέτρους, αριθμό καναλιών κτλ. Κάποιες χώρες δεν έχουν υιοθετήσει κανέναν κανόνα. Η το περίπλοκο παζλ που έχει δημιουργηθεί λόγω των πολλών και διαφορετικών εθνικών κανονισμών δεν επιτρέπει να εγκαθίστανται εύκολα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια άλλη χώρα και να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Αυτές οι διαφορές θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ακριβώς παρεμποδίζοντας ε, το δικαίωμα εγκατάστασης ε, και ελευθερίας κίνησης των υπηρεσιών. Δεν πρέπει να υπάρχει ελευθερία διακίνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη στην, στην, αρχή, ε, ε, στην αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων ακριβώς δείχνει ότι πιστεύει ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε πολλά κράτη-μέλη απέδειξαν ότι ο στόχος της οδηγίας είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς και εσωτερικής περιοχής χωρίς ε, σύνορα για τα οπτικοακουστικά μέσα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ένα ε, και την προστασία των ε, στόχων ε, και των ενδιαφερόντων του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό ακριβώς, κατά την άποψή μου, ο βασικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίσει την ελευθερία και τον πλουραλισμό και θα πρέπει να παίξει ένα πιο δραστήριο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο των αγορών των ΜΜΕ. Επομένως, όπως και αν ονομαστεί η μελλοντική οδηγία, δεν έχει σημασία, θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες ρήτρε διασφάλισης και για τους στόχους γενικού ενδιαφέροντος, γενικού συμφέροντος, διότι η σημασία τους ήδη ε, αναφέρεται και ε, τονίζεται στα εκτιμώντας που δεν εντάσσονται όμως μέχρι στιγμής στον συντονισμένο τομέα. Ο Ευρωπαίος ο νομοθέτης πρέπει να σεβαστεί βέβαια και την αρχή της επικουρικότητας, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το άρθρο 51 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που λέει ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και να προωθήσουμε την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων, που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Χάρτας. Σε πολλές περιπτώσεις ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε με βάση το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης, που είναι το αντίστοιχο άρθρο του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Χάρτας, ότι το κράτος δεν είναι ο, ο εχθρός, αλλά ε, είναι αυτός ο οποίος θα διασφαλίσει την ελευθερία και τον σεβασμό των, της νομοθεσίας και του χάρτη. Με βάση την νομολογία του δικαστηρίου και με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί διαφορετικά standards έχουν υιοθετηθεί, εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα πρότυπα όταν υιοθετεί μέτρα για την πρόθεση της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες μέσω μαζικής ενημέρωσης. Με τη μορφή ελάχιστων ε, ε, προτύπων, προδιαγραφών που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη με τα αντίστοιχα και ανάλογα μέτρα. Η οδηγία, όσο έχει τώρα, δεν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τέτοιου είδου νομοθεσία στους συντονισμένους τομείς. Για να ολοκληρώσω, εάν η εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα μέσα μεσικής ενημέρωσης μπορεί να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό πολίτη από το να αντιμετωπίσει με, κοινές, σκηνές σεξ στην ε, τηλεόραση στις 4 η ώρα το απόγευμα, γιατί να μην μπορεί ο ίδιος πολίτης να προστατευτεί από το να βλέπει περιεχόμενο το οποίο ε, τον επηρεάζει με άσχημο τρόπο τις, τα οικονομικά και τα πολιτικά του συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Προχωρούμε τώρα στο δεύτερο μέλος του πάνελ που είναι ο κύριος Μάριος Ντράγκομιρ μάνατζερ του προγράμματος χαρτογράφησης ψηφιακών μέσων και την κυρία Μαγδά Βόλτερ, η οποία είναι περιφερειακή συντάκτης. Ο κύριος Ντράγκορμιρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε τα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος ε, τα οποία τρέχουν εδώ και τέσσερα χρόνια από τον οργανισμό μας που είναι η ε, Ανοιχτή Κοινωνία, ε, το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας, Open Society Foundations. Καλύπτουμε μέση, μέσα ενημέρωσης διεθνώς, αλλά τα τελευταία χρόνια ασχοληθήκαμε με την έρευνα και την ε, ακολουθούμενη πολιτική. Ε, ε, τα στοιχεία που έχουμε προέρχονται από τα ψηφιακά μέσα, από τη χαρτογράφηση ψηφιακών μέσων, όπως σας είπα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, τα περισσότερα, περισσότερα από τα μισά προγράμματα έχουν δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμα. Είναι αυτού του είδους όπως κρατάω στα χέρια μας και τα βρίσκεται και στο διαδίκτυο. Είναι όλα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. 13 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλική, η Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, ε, η Σουηδία και το Ενωμένο Βασίλειο. Ε, αυτές οι εκθέσει είναι διαθέσιμε. Ε, και επίσης για υποψήφιες χώρες και δεχόμενα υποψήφιες χώρες έχουν δημοσιευθεί Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κροατία, Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία. Σήμερα θα καλύψουμε. Ε, είχαμε ορισμένες διαφάνειες, αλλά ε, ε, συνεχίζω την ομιλία μου καλύπτουμε τρία θέματα για τη σημερινή συζήτηση και η βασική, <laughs> να, εδώ είναι οι διαφάνειες. Έχουμε λοιπόν καλύψει 60 χώρες από τη Λατινική Αμερική όπως βλέπετε, την Βόρεια, την, τις Ηνωμένες χώρες στην Αφρική. Αλλά όπως σας είπα η βασική μας εστίαση είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, 24 ευρωπαϊκές χώρες έχουμε καλύψει. Σήμερα θα παρουσιάζουμε λοιπόν ακριβώς αυτές ε, τα ευρήματα τα που έχουμε για την ιδιοκτησία, το θέμα της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωση και συνάδελφός μου η Μάγδα θα σας παρουσιάσω ορισμένε συστάσεις που προέκυψαν από αυτό το έργο. Ε, αυτές ε, οι εκθέσεις έχουν συνταχθεί από ανεξάρτητους τοπικούς εμπειρογνώμονες και έχουν ελεγχθεί από ένα μεγάλο αριθμό συντακτών. Όταν μιλάμε για καθεστώς ιδιοκτησίας, ορισμένα από τα στοιχεία που διαπιστώσαμε σε αυτές τις χώρες και βασικά ασχοληθήκαμε με την ψηφιοποίηση και τα ψηφιακά μέσα, ε, πολυμορφία και πρόσβαση και ένα από τα στοιχεία που διαπιστώσαμε είναι ενισχυμένη συγκέντρωση ε, ιδιοκτησίας τα επίπεδα συγκέντρωση της ιδιοκτησίας ε, ήταν ήδη υψηλά, μη επιτρέποντας και πιστεύαμε, ε, και μη επιτρέποντας περαιτέρω διόγκωση της ε, πυκνότητας αυτής της ιδιοκτησίας. Όμως διαπιστώσαμε και απορρίθμιση των κανόνων ιδιοκτησίας, ιδίως όταν πρόκειται για συνειδιοκτησία. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένες, ε, ορισμένα ποσοστά λαθών στις ε, έρευνες τις οποίες κάναμε και επίσης διαπιστώσαμε στην Ολλανδία, στη Σλοβενία και στη Ρουμανία επήλθε μία απορρίσμηση του, των κανόνων ιδιοκτησίας. Βεβαίως το βασικό μας ενδιαφέρον ήταν η ανεξαρτησία της σύνταξης. Ε, πολλοί ερευνητές αυτού του τομέα ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ακριβώς τη διασύνδεση μεταξύ της ε, συγκέντρωσης ε, εξουσίας, ιδιοκτησίας αν θέλετε και ανεξαρτησίας της δημοσιογραφίας η, η πολιτική ελίτ, η, σχίουσα, η άρχουσα τάξη της πολιτικής και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενομέρωσης έχουν συνδεθεί ακόμα πιο στενά στην εποχή μας, παραδείγματος χάρη ε, στη ε, Σλοβενία, σε άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης έχουν στενότατες σχέσεις και επαφές και κοσμικές επαφές με πολιτικούς, κυβερνήσεις κλπ. Ε, όσον αφορά τώρα τη δημοσιογραφία, αυτοί, αυτές οι στενές ε, διασυνδέσεις έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο βλάψει την ουδετερότητα των ε, ειδήσεων. Όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ισχύ της ψηφιοποίησης και την αναδιάσωση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο συμβαίνει ότι είναι ότι η αναδιάρθρωση επιταχύνεται ε, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους ε, και ο ορθολογισμός. Η Λιθουανία πρόσφατα στη Λιθουανία ε, μια κύρια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας δηλαδή απέλησε το 1 τέταρτο των δημοσιογράφων. Αυτό βλάπτει ιδιαίτερα την ερευνητική δημοσιογραφία την οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε σήμερα διότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι το αίμα, είναι η καρδιά της δημοσιογραφίας και βεβαίως έχει μειώσει επίσης τη δέσμευση των εκδοτών να υποστηρίξουν ένα, μια δημοσιογραφία η οποία ενέχει κινδύνους, ενέχει ρίσκο. Ε, εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε την επιβίωση του ερευνητική, της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Έχουν επίσης υιοθετηθεί ε, νόμοι για την συκοφαντία και για την ε, ιδιωτικότητα, οι οποίοι δημιουργούν προσκόμματα στην ελεύθερη δημοσιογραφία. Ρύθμιση Βλέπουμε συνεχείς συμβιβασμούς αλλά και παραντάσεις πολλών κυβερνήσεων σε, αυτές τις, σε πολλές χώρες ε, ε, και μάλιστα περιορισμό της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν μόνο περιφερειακές αρχές. Μία τέτοια αποπτική αρχή, το οπτικοακουστικό, η οπτικοακουστική ρυθμιστική αρχή στο, του Ναβάρο ε, έκλεισε καταργήθηκε φέτο. Επίσης διαπιστώσαμε πριν από 6-7 χρόνια από τη μελέτη μας υπάρχει ένα οξύ πρόβλημα στην κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή αυξανόμενη πολιτικοποίηση που διώχνει τους ακροατές ή τους αναγνώστες. Ε, επίσης, ε, ε, ένα άλλο γεγονός που διαπιστώσαμε είναι κυβερνητική διαφήμιση. Πάρα πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα κονδύλια τους για την στήριξη φιλικών ε, προς, αυτές, ε, ε, προς αυτούς μέσα ενημέρωσης, χρηματοδοτούν δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης που είναι φιλικά προσχήματα προς την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Πράγματι αυτό είναι μια μακρά παράδοση και έτσι επηρεάζονται από την πολιτική εξουσία τα μέσα ενημέρωσης δεν γίνεται άμεση χρηματοδότηση αλλά μέσω εταιρεών και ιδρυμάτων. Έτσι λοιπόν και στη Σλοβενία υπάρχουν ε, κρατικές εταιρείε οι οποίες έχουν αποστείλει τις διαφημίσεις τους. Άρα λοιπόν αυτή η ενίσχυση, η, η, η απόσταση ε, πιστώσεων για διαφημίσεις σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης έχει αρνητικά αποτελέσματα ε, πολλές φορές βεβαίω ως δικαιολογία λένε ότι είναι το κλίμα λιτότητος, η έλλειψη πιστώσεων κλπ. Όμως παραμένει γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική επιρροή μέσω της ε, διοχέτευσης ε, κρατικών διαφημίσεων, κρατικών τρόπων προώθησης, προαγωγής. Συστάσεις, η Μάγδα. Ευχαριστώ πρόεδρε πριν αναφέρω τις ε, βασικές συστάσεις που προέκυψαν από την ε, χαρτογράφηση ψηφιακών μέσων και από την ανασκόπηση των ευρωπαϊκών χωρών, την έκθεση δηλαδή αυτή που πρόσφατα εκδώσαμε και που βάλαμε στην Επιτροπή, θέλω να κάνω δύο-τρεις γενικές παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτές οι συστάσεις δεν είναι συστάσεις του Ιδρύματος Ανοιχτής Κοινωνίας, Open Society. Είναι συστάσεις που βασίζονται στην ανάλυση του, της, των εκθέσεων που έχουμε κάνει ανά χώρα, όπως είπε ο συνάδελφός μας. Οι περισσότερες αυτές ε, εθνικές εκθέσεις ε, περιέχουν συστάσεις για κάθε χώρα. Άρα, οι συστάσεις τις οποίες θα αναφέρω εγώ αποτελούν το συγκερασμό όλων αυτών των συμπερασμάτων που υπάρχουν στις εκθέσεις και οι οποίες συστάσεις έχουν επιβεβαιωθεί και εγκριθεί από διάφορες συζητήσεις τραπέζης που έγιναν με στόχο να συγκεραστούν οι εθνικές συστάσεις. Βάσει αυτών που είπαμε σήμερα, πιστεύω ότι αυτά που προτείνουμε και αυτά που πιστεύουμε ε, είναι ορισμένα ελάχιστα πρότυπα για να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες επιπτώσεις και όπως εκφράστηκαν ανησυχίες πολλών μελών εδώ, ε, ιδίως στο σημερινό κλίμα πολλών κρατών μελών ε, και να αντιμετωπίσουν επίσης και το θέμα της υπερβολικής ρύθμισης. Όταν υπάρχουν μήνυμου πρότυπα πρέπει να αποφευθεί, μπορεί να αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος. Καταρχάς το θέμα της ιδιοκτησίας. Ε, αυτό είναι προτείνουμε όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ελάχιστα πρότυμα για τις νομικές διατάξεις και μηχανισμούς που θα ε, αποφύγουν που θα, ε, την, την πολιτική επιρροή στα μέσα, ε, στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και θα διασφαλίσουν διαφάνεια της ιδιοκτησίας. Επίση, πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ερμονίσει τους κανόνες ιδιοκτησία μέσων ενημέρωση. να αλλάξει ή ανανεώσει το AVMSD. Ε, είναι ο πιο δύσκολος στόχος αυτός βεβαίως, αλλά εμείς προτείνουμε και πάλι αυτό είναι ένα ελάχιστο επίπεδο ε, να ε, βρεθούν νέα μοντέλα ε, τα οποία θα ρυθμίζουν τον, τα μέσα μέσα και ιδίω στην οπτικοακουστική πτυχή μέσω της οδηγίας αυτής της Κομισιόν. τώρα, για τους δημοσιογράφους, τη δημοσιογραφία. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρεμβάσεις ε, από, ε, την από κυβερνήσεις. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ακολουθήσει ε, την πρωτοβουλία α, να, να, ακολουθήσει την πρωτοβουλία αποκατάργησης κατάργησης της πολιτικής σκοπιμότητας και της πολιτικής εξάρτησης ε, των ιδιοκτητών στα μέσα ενημέρωσης, να επίσης να ε, υιοθετήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια και σε διαδικασίες για την προβολή, την κρατική προβολή στα μέσα ενημέρωσης, προ, κρατική προβολή και διαφήμιση. Υπάρχουν ήδη ε, περιφερειακά, περιφερειακοί μηχανισμοί, περιφερειακοί μέθοδοι ε, που επιβάλλουν κανόνες για αυτή την ε, διαφήμιση και επίσης υπάρχει και η αντίστοιχη πρωτοβουλία πέραν του Ατλαντικού από την ε, Αμερικανική ε, Πρωτοβουλία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτό τον τρόπο προβολής και διαφήμισης. Επίσης προτείνουμε να υποστηριχθεί, να ενισχυθεί ένα πλαίσιο ευθύνης ε, και ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό είναι επίγον δεδομένου ότι ε, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία υλοποίησης αυτών των συστάσεων είναι ε, ε, εμφανές πόσο μοιάζουν οι δικές μας συστάσεις με τις συστάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και στο σχέδιο έκθεσης που έχουμε δει ε, επιβεβαιώνονται οι αρχές μας, επιβεβαιώνεται ο, ο, παραλληλισμός των αρχών μας και μειότητα των αρχών μας μεταξύ του δικού μας οργανισμού και της Επιτροπής σας, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ο κύριος Ράσταλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και κυρία την κυρία Βέμπερ για την ευκαιρία που μας δίνεται να μπούμε στην καρδιά της ελευθεροτυπίας ε, και της πολυφωνίας του τύπου. Να σας πω εγώ ότι εκπροσωπώ την Ένωση Εκδοτών ε, εφημερίδων. Είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση διεθνής και εκπροσωπούμε πάνω από 5.200 εθνικές, τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες που εκδίδονται στα περισσότερα κράτη-μέλη, Νορβηγία, Επαιτία και Σερβία. Γίνεται σε κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο μας αυτή η ακρόαση. Δεν θα σας εκπλήξει ότι ε, όλοι μπορούν να επιλέξουν σήμερα από τεράστια ροή και γραπτή ενημέρωσης και ψηφιακής. Και όλοι οι εκδότες ψάχνουν νέα μοντέλα επιχειρηματικά για να φύγουν, να ξεφύγουν από το χθεσινό γραπτό ε, περιβάλλον στο αυριανό ψηφιακό. Ωστόσο, οι προκλήσει ε, είναι ίδιες. Εμείς θέλουμε να δίνουμε στους χρήστε και στους αναγνώστες έγκυρες πληροφορίε από όλες τις πλατφόρμες για ταμπλέτες, τα ε, ψηφιακά και στι χιλιάδες ε, κλασικές εφημερίδες. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε το ζωτικό μας ρόλο και να διευκολύνουμε τι ανοιχτέ και ειλικρινεί συζητήσει. Τι χρειάζεται τώρα ο εκδοτικό κόσμος για να συνεχίσει να δημιουργεί σε αυτό το κλάδο της οικονομίας. Τι ζητάμε από εσά, τους νομοθέτες μας. Πέντε σύντομα σημεία θα ήθελα να σας αναφέρω. Πρώτον, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα που τα κράτη-μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα. Σύμφωνα με τη συνθήκη, όπως ακούσαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στη ρύθμιση της πολυφωνίας του τύπου, μόνο δια του ανταγωνισμού. Και υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί λόγοι είναι πολύ διαφορετική αγορά του τύπου από χώρα σε χώρα για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και η κατανάλωση εντό εισαγωγικών τύπου διαφέρει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Και το θέμα της πολυφωνίας του τύπου μπορούν να το ρυθμίσουν μόνο εθνικές αρχές που ε, προσαρμόζουν τα πράγματα με βάση τις τοπικές, εθνικές και περιφερειακές τους ε, πραγματικότητες. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντική η αυθορύθμιση. Έχουν ε, εγκριθεί κώδικες εντολογίας από διάφορους κλάδους, συχνά σε συνεργασία με δημοσιογράφου ή και από μεμονωμένε εφημερίδε. Υπάρχουν εφημερίδε που έχουν τον ίδιο του το διαμεσολαβητή, όπω είναι η Guardia στη Βρετανία ή η η ελπαις στην Ισπανία. Ε, υπάρχουν ε, επίσης ε, και ε, μεγάλες διαδικασίες. Οι ανεξάρτητες ε, αρχές και οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι γνωρίζουν τι ισχύει στη χώρα τους. Λοιπόν, κάθε χώρα ξέρει πάρα πολύ καλά ε, τι συμβαίνει και αυτό δεν υπονομεύει την ελευθεροτυπία. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπερασπιστώ την αξιόπινη συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων που πάντα θα διώκεται ποινικά. Εδώ είναι πολύ σημαντικό επίσης για όλους, αναγνώστες, εκδότες και πολιτικούς, να αναγνωρίσουν το ρόλο ε, του αρχισυντάκτη. Ο αρχισυντάκτης φέρει ε, ακέραια την ευθύνη για την ε, συντακτική γραμμή και την καθημερινή έκδοση της εφημερίδας και ασφαλίζει και την ισορροπία των γνωμών και των απόψεων. Είναι σημαντικό να έχουμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη τα μάτια των αναγνωστών. Αν χάσει ο αναγνώστης την εμπιστοσύνη σε μια εφημερίδα θα στραφεί σε ε, άλλη μορφή ενημέρωσης. Και αυτό είναι ο νόμος τελικά της ζήτησης και της προσφοράς. Ε, και αυτό είναι καλύτερο από οποιοδήποτε νομοθετικό μέτρο. Γιατί η μόνη βάση για ένα σοβαρό μέσο ενημέρωσης είναι η εμπιστοσύνη του αναγνώστη ή του χρήστη. Και αυτή είναι και η απάντηση στο δίλημα που έφερε ξεότιμο μέλος από τη Ρουμανία ότι υπάρχει ελευθερία και έλλειψη ελευθερίας ε, στις εκδόσεις. Ε, θέλω να αναφερθώ και στο ιδιοκτικό κτησιακό καθεστώς. Η συγκέντρωση ε, στα χέρια ε, κάποιου ε, δεν έχει να κάνει με την πολυφωνία. Το θέμα δεν είναι ποιο είναι ιδιοκτήτη, αλλά αν υπάρχει αρκετό ανταγωνισμό. Αυτό ε, θα πρέπει να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, ακριβώ σε πλαίσια όμω ανταγωνισμού, για να υπάρχει ένα περιβάλλον να μπορούν να εργάζονται όλοι. Υπάρχουν εφημερίδε ε, και μίντια που κάθε μέρα υποφελούνται από το γεγονό ότι ανήκουν σε ένα μεγάλο όμιλο. Και κατά τη διάρκεια αυτή τη κρίση του επέτρεψε να είναι πιο ανθεκτικά. Θα είχαν κλείσει πολλέ εφημερίδε πρόσφατα, αν δεν ανήκαν σε ένα μεγάλο όμιλο, σε μια μεγαλύτερη δομή μηντιακή. Ταυτόχρονα συμφωνώ τους με εκείνους που ε, προλαλήσαντες που είπαν ότι υπάρχει ανάγκη διαφάνεια στα ιδιοκτησιακά και στα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτικών. Προφανώς αυτό είναι τα θεμέλια για οποιοδήποτε τομέα και πόσο μάλλον για τον τύπο. Στη συνέχεια, οποιαδήποτε αξιολόγηση, εκτίμηση της πολυφωνίας του τύπου δεν θα πρέπει να εξετάζει μόνο τα κλασικά μέσα ενημέρωσης. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν μεγάλες τεχνολογικές πολυεθνικές εταιρείες, γίγαντες μη Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο που έχουν τεράστια επίπτωση ε, στο πώς ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει παρακαλώ να τα κοιτάξετε αυτά ε, προσεκτικά. Υπάρχουν πλατφόρμες που συγκεντρώνουν ειδήσει και εκμεταλλεύονται αυτές για τους δικούς τους εμπορικούς σκοπούς ε, και χωρίς καμία μορφή συνένεσης υπάρχει και θέμα βέβαια εδώ πνευματικών δικαιωμάτων και copyright. Και τέλος, αυτό είναι αυτονόητο και προφανέ ότι για να είναι πλήρως ανεξάρτητε οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωση θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα. Οποιοδήποτε περαιτέρω περιορισμοί, απαγορεύσει διαφημίσεων να αποφευθούν γιατί αυτό επηρεάζουν την ελευθερία του τύπου. Επίσης θέλουμε και την υποστήριξή σας για να πέσει ΦΠΑ. Ε, για να εξισωθούν ε, με ε, το ΦΠΑ για τον τύπο. Εμείς πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε νομοθετικά μέτρα που ε, φιλοδοξούν να θέσουν εντό εισαγωγικών πρότυπα και προδιαγραφές για την ελευθερία του τύπου, το μόνο που κάνει είναι να περιορίζει την ελευθεροτυπία. Ο νομοθέτης θα μπορούσε ή θα ε, έπρεπε να ορίσει ε, ηθικά στάνταρ και ε, όμως αυτή δεν πρέπει να ρυθμίζεται νομοθετικά, δεν έχει να κάνει και δεν έχει καμία σχέση με την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ευαίσθητες καταστάσεις σε εθνικές ε, πραγματικότητε σε διάφορα κράτη-μέλη, μάλιστα όπω ακούσαμε προηγουμένω. Αλλά οι Εφημερίδε και τα μέσα ενημέρωσης ιδιοσογραφίας θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν μόνοι του και να εργάζονται ε, εντό του συντάγματο, των ρυθμιστικών ε, ε, αρχών και του ποινικού δικαίου των κρατών μελών του. Οι νομοθέτε τι δουλειά έχουν ε, να προάγουν την ελεύθερη ε, συζήτηση στα κράτη-μέλη με πολιτικές για την τόνωση του τύπου, του ανεξάρτητου τύπου, του αξιόπιστου τύπου, ε, όπως έχει κάθε δικαίωμα ο πολίτης να ενημερώνεται. Πράγμα που συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη για να αυξηθεί η πολυφωνία και η ελευθερία του τύπου. Όσο καλόβουλες και να είναι οι προθέσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία για προδιαγραφές και πρότυπα κινδυνεύει ε, πάρα πολύ να υπονομεύσει και να βλάψει και την ελευθερία. Η ελευθερία του τύπου θα είναι πάντα η εγγύηση της πολυφωνίας και ε, της ενημέρωσης στις δημοκρατικές κοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράσδαλ. Τώρα ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα χρόνου ε, στις 12.30 θα πρέπει να έχουμε τελειώσει διότι συνεδριάζουν οι συντονιστές και έχει και μεγάλη ημερήσια διάταξη. Και θα έχουμε και τη ε, Γενική Διευθύντρια. Λοιπόν, παρακαλώ να περάσουμε αμέσω στο επόμενο πάνελ, να αλλάξουν οι ομιλητές στην έδρα και μετά θα κάνουμε συζήτηση και για τα δύο μαζί. Έτσι, κοινή. Για τα δύο πάνελ. Το παρόν και το επόμενο. θα είναι και το τελευταίο. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα μπορέσετε να απαντήσετε σε λίγους ερωτήσεις. If the third round of panelists are kind enough... Λοιπόν, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, οι ομιλητές του τρίτου πάνελ να έρθετε. Παρακαλώ. The third round of panelists is going to be... Έχουμε τον κύριο Άρνε Κόνικ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Καλώς ορίσατε. Mr. Ο κύριος Ολιβιέ Μπαζίλ από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και ο κύριος Βίλιαμ Χόσλεϊ που εκπροσωπεί το Σύνδεσμο των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Είστε παρόντες όλοι. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, σκεφτείτε και το χρόνο παρακαλώ για να τελειώσουμε στις 12.30. Ο κ. Άρνε Κιόνικ. Από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Μιλάμε για βασικά ερωτήματα και χαίρομαι που μπορούμε εδώ να απευθυνθούμε και σε πολιτικούς, διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και έλλειψη πολιτικής θέλησης. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που χαιρόμαστε που είμαστε εδώ είναι αυτός. Πολλά ε, χρόνια τα πέρασα στην Τουρκία και ε, έχουμε 90 οργανώσεις που συμμετέχουν σε μία προσπάθεια για να ελευθερωθούν οι φυλακισμένοι δημοσιογράφοι. Στην Τουρκία υπάρχει έλλειψη ελευθερίας του, του τύπου, έλλειψη αξιοπιστίας, δεν υπάρχει διάλογος ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τους εργα, εργα, εργοδότες, ε, πιέσεις στα συνδικάτα, πιέσεις από την κυβέρνηση και ε, ε, αυτό, όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα 80 ε, δημοσιογράφοι να είναι φυλακισμένοι. Και η Τουρκία είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων. Η ελευθερία των ΜΜΕ είναι κάτι ευρύτερο από αυτό που ανέφερε, αναφέρει η κυρία Βέμπερ στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Εμείς ε, είμαστε παρόντες ε, πολλά χρόνια και προσπαθούμε να πετύχουμε αυτή την ελευθερία, γι' αυτό καλωσορίζουμε και την πρωτοβουλία της κυρίας Βέμπερ. Ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνας. Η ελευθερία των μέσων ΜΜΕ και του πλουραλισμού είναι θεμελιώδει ελευθερίες, τις οποίε πρέπει να διαφυλάξουμε Δεν θα εκπλήξει κανέναν σας εδώ το ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα παραβίασης της ελευθερίας των, του τύπου στην Ευρώπη, στην Λευκορωσία και σε άλλα μέρη. Ε, υπάρχει παραβίαση από, πολλές, από πολλούς κρατικούς φορείς ε, χωρίς να επιβάλλονται ε, οι, ε, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση, να διαμαρτυρηθούμε τουλάχιστον. Ε, υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες οι οποίες επηρεάζουν ε, και την ελευθερία των δημοσιογράφων. Τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν ε, πριν από μερικά χρόνια την διακήρυξη του Ρέκεβικ που, λέει, που έλεγε ότι υπάρχει λόγω της 11 η Σεπτεμβρίου μια υπερβολή, ένας υπερβολικός περιορισμός του τύπου το ίδιο έχει να κάνει και με την, ε, ε, και την, τα ηλεκτρονικά μέσα και τις ηλεκτρονικές πληροφορίες όσον αφορά τις πηγές, ε, η, το δικαίωμα φωτογράφησης. Η πολιτική παρέμβαση είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα όταν έχουμε χώρες όπου η πολιτική ε, ελέγχουν ε, τις πολιτικές πληροφορίες, ε, τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στις πολιτικές συγκεντρώσεις κτλ. Ο δημοσιογράφος, η δημοσιογραφία αναφέρεται σαν η πέμπτη εξουσία πολλές φορές. Όμως για μας δεν έχει τόσο σημασία η εξουσία όσο η πληροφόρηση. Δεν είναι θέμα εξουσίας, είναι, γενικά, είναι δημόσιο αγαθό η δημοσιογραφία πιστεύουμε εμείς. Γι' αυτό απευθύνουμε μια έκκληση στις ευρωπαϊκές αρχές αλλά και στις ε, εθνικές αρχές ε, έτσι ώστε να αναφερθεί αυτός ο βασικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να τονιστεί ακριβώς η, σημασία της ελευθερίας ε, του τύπου. Γι' αυτό εδώ έχουμε, πρέπει να δούμε και την ισορροπία ανάμεσα στα δημόσια και στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών για τον πλουραλισμό των ΜΜΕ η οποία έγινε ε, θετικά από, την, ε, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πολλοί δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν σε ποιον ανήκει η, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στον τομέα αυτό. Και θα, όταν συζητάμε για την ε, ιδιοκτησία των αγαθών θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ένα βασικό ερώτημα. Ποιο θα πληρώσει για τον, ε, την δημοσιογραφία στο μέλλον. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, αλλά όλη την κοινωνία εν γέννη. Η ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι ε, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Και χαιρόμαστε γιατί το σχέδιο αυτό α, ε, της έκθεσης το λαμβάνει υπόψη. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ε, και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ασχολούμεθα με αυτό καθημερινά. Θέλαμε να σας πούμε ότι οι πολιτικές ασφάλειας αναφέρονται και στην ατιμορρησία. Δεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες αρχές ε, να παραβιάζουν την νομοθεσία, να, παραβιάζουν, να πιέζουν, να ασκούν πιέσεις ε, και να ε, δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα χωρίς ε, να υπάρχει μία απάντηση. Εδώ μιλάμε για τα πολε... τα, όταν μιλάμε για πολεμικά εγκλήματα, εκεί υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαστήρια τα οποία ασχολούνται με αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μιλάμε τώρα και για τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων. Υπάρχει και μια δήλωση που αφορά περισσότερο, μια διακήρυξη που αφορά περισσότερο τις εμπόλεμες περιπτώσεις, αλλά θα μπορούσε να αφορά και τους δημοσιογράφους σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολλοί δημοσιογράφοι ασχολούνται με την ελευθερία και τον πλουραλισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι συμμετέχουν ενεργά οι οργανώσεις δημοσιογράφων καταδικάζουν πολλές φορές ε, την, ε, ε, την εμπορική εκμετάλλευση των, της δημοσιογραφίας και βλέπουμε ότι έχουμε μια εμφανή παρέμβαση των χορηγών στην κυκλοφορία της, της πληροφορίας ή στο δικαίωμα να λαμβάνονται φωτογραφίες στην, ε, στο σχέδιο έκθεσης ε, των, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρονται όλα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να σεβαστούμε και την αναθεωρημένο χάρτη κοινωνικών δικαιωμάτων της Ευρώπης. η δυνατότητα κάλυψης ε, συλλογικών ε, συμβάσεων θα πρέπει να ισχύει για όλους, ε, ακόμα και αν εργάζονται για μικρές επιχειρήσεις για, ή απασχολούνται με μερική απασχόληση. Στον τομέα δυστυχώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι επισφαλής η η σύμβαση, το εργασιακό μάλλον καθεστώς των δημοσιογράφων. Εκτός όμως από, την, από το εργασιακό καθεστώς, από τους μισθούς και τα λοιπά, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις συνθήκες εργασίας και θα πρέπει να εκφράζονται συλλογικά και δημοσιογράφοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Υπάρχει και ο ρόλος των κανονιστικών οργάνων που θα πρέπει να εξετάσουμε και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα κανονιστικά καθεστώτα που ισχύουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται άλλοι τομείς γιατί μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές ε, ερμηνείες. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο να ισχύει σε όλους. Ε, Παραδείγματο χάρη αυτό το οποίο έγινε στην Ουγγαρία για την αρχή ε, τύπου, έτσι όπως έχει διαμορφώθηκε άσχημα κατά την άποψή μας. Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε τον σοβαρό αντίκτυπο που έχει η κρίση στον τομέα. Είναι διτή, διτός ο αντίκτυπος. Υπάρχει η κρίση αυτή καθεαυτή και ε, η κρίση έτσι όπως την εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες για να αυξήσουν ε, το περιθώριο κέρδους τους. Εμείς ε, εδώ και χρόνια προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την, την κρίση γιατί τα τελευταία τρία χρόνια χιλιάδες δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους ή συνέχισαν να, δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Αυτή τη στιγμή πλήττεται η Πορτογαλία. Ποιος θα αγοράσει ένα χρεοκοπημένο τηλεοπτικό κανάλι. Ένα τρίτο, το 1 τρίτο του, του, του, του, της έγκυρης εφημερίδας Ελπαΐ στην Ισπανία απολύεται. Ε, αντίστοιχα συμβαίνουν και στην Νορβηγία. Ε, επίσης ε, το BBC και η France Television περιορίζουν τις δαπάνες τους, ε, πολλά περιοδικά κλείνουν σε όλη την Ευρώπη και το θέμα δεν είναι θέσεις απασχόλησης, είναι, είναι θέμα δημοσιογραφίας, είναι θέμα δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών να ενημερώνονται σωστά. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε έγκυρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση. Η δημοσιογραφία δεν είναι απλώς ε, μια απασχόληση, είναι και θέμα ε, κοινωνίας. Πολλοί δημοσιογράφοι ζουν ε, βέβαια σε περιβάλλοντα διαφθοράς φτώχειας. Όμως Δεν μπορούμε να ε, παραβιάζουμε την ελευθερία του τύπου. Ε, χτες, η 5η Νοεμβρίου, ήταν η ημέρα της, του ανεξάρτητου δημοσιογράφου. Και ε, ζητήσαμε από όλα τα μέλη μας να εορτάσουν αυτή την ημέρα. Και αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε τους Τούρκους συναδέλφους ε, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό για την κατάσταση στην Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε υπόψη την πίεση χρόνου δεδομένου ότι θα συγκεράσουμε και τις δύο συζητήσεις και του προηγούμενου πάνελ και του τελευταίου και προχωρούμε στον κύριο Ολιβίε Μπαζίλ από τους Reporters Χωρίς Σύνορα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα περιορίσω την τοποθέτησή μου, διότι πραγματικά μας ενδιαφέρει να κάνουμε ανταλλαγή απόψε μαζί σας. Βέβαια, εξ ονόματος των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα απευθύνομαι σε εσά, αλλά κυρίως βάσει του δικτύου Ζαχάροφ, γιατί έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με τους βραβευθέντες στο βραβείο Ζαχάροφ την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου και συμμερίζονται τις δικές μας ανησυχίες και συμφωνούν για να σας πούμε από κοινού τα εξή. Από το 2008 η κατάσταση της ελευθεροτυπίας στα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, δεν έχει σταματήσει να ε, ε, μειώνεται και Έχουμε δημιουργήσει και ειδικό γραφείο για να μελετάει αυτά τα θέματα και για την πολιτική ε, γειτονίας. Ε, η μεγαλύτερη απειλή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι νομοθετική. Δηλαδή, εδώ και τέσσερα χρόνια βλέπουμε να αναβιώνουν μια σειρά μέτρων νομοθετικών ή κυβερνητικών. Το ξέρω ότι είναι εθνική αυτή η υπόθεση και κρατών μελών, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα κράτος που να μην υποχωρεί υπόθεση τη ελευθερίας έκφραση, της ενημέρωση και του τύπου. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν θα σας μιλήσω για την Ουγγαρία, δεν θα σας προσβάλλω. Τα γνωρίζετε αυτά πολύ καλά. Αλλά ε, ε, τα η ε, Ουγγαρία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Ιταλία, ε, έχουν γνωρίσει αντίστοιχα προβλήματα χωρίς να υδρώσει ε, το αυτή κανενός στην Ευρώπη ε, και έχουν παραπιαστεί τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει παράδεισος για όλο τον κόσμο. Μπορεί να έρθει ε, όποιος θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διώξει ε, χειριστικά δημοσιογράφους. Η Ένωση υποτίθεται πολεμά κάποια ε, κράτη που θέλουν να επιστρέψουμε στο να διώκεται ποινικά η βλασφημία στην Ιρλανδία έχει πρόστιμο 25.000 και η Μάλτα διώκει τα θέματα βλασφημίας. Στο Βέλγιο που είναι πολύ καλό κράτος σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών το Βέλγιο λοιπόν εγκρίνει ε, μάλλον έχει μια πολιτική στο γαλλόφωνο τύπο ένα είδος υγειονομικού κλειού. Υπάρχουν ε, κόμματα που αποκλείονται από τη δημόσια συζήτηση. Ενώ ε, στη Φλάνδρα ο ίδιος νόμος οργανώνει αυτή την κατάσταση. Και τελικά είναι σχιζοφρενείς οι συνθήκες που επικρατούν. Γιατί τα λέω αυτά. Διότι ως διεθνής οργάνωση βλέπουμε χώρες πάρα πολύ ελευθεριοκτόνες. Πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ενώ τώρα έχουμε τεράστιες αντιφάσεις στην Ένωση σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και είναι πολύ δύσκολο ε, να ε, δακτυλοδεικτούμε ε, κάποιες χώρες που είναι πιο προχωρημένες πολλές φορές από ορισμένα κράτη-μέλη στα κείμενα των νομοθετικά, όχι στις αξίες και ε, ε, αυξάνονται και οι δίκες με τις ε, νομοθετικές υπερβολές και οι διαδικασίες που είναι η μεγάλη αγάπη πλέον μια μεγάλη πολιτική τάξη από όλα τα κόμματα που κάνουν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και πίσω από αυτά τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους. Ακούσαμε σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης τι συμβαίνει. Η μεγαλύτερη κατηγορία των δημοσιογράφων είναι αυτή και είναι πάρα πολύ εύθραυση η κατάσταση. Αυξάνονται γίνονται φαινόμενα ε, ε, ε, αυτολογοκρισίας και οι ελεύθεροι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν δίκες 2, 3 και 5 με πρόστιμα 10.000 ευρώ για να μην μιλήσουμε για ποινές φυλάκισης που εμφανίζονται όλο και περισσότερο στα νομοσχέδια ενώ εμείς θέλουμε να αποποινικοποιούνται τα λεγόμενα εγκλήματα τύπου. Έχουμε προβλήματα και με τους πολιτικούς σήμερα, με τη στάση τους. Δεν μιλώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ε, για τα εθνικά κοινοβούλια, για την αντίληψη που έχουν για τα μέσα ενημέρωσης, ε, ο λόγος, ε, ποιος είναι και τι λένε, να οργανωθεί ο τύπος, να υπάρχει ισορροπία, να λαμβάνεται υπόψη, το ακούσαμε και σήμερα, η λεγόμενη αποτυχία της αυτορύθμισης και ότι πλέον χρειάζεται να τα αναλάβει αυτό κάποιος άλλος φορέας. Και ε, πολύ συχνά αυτό διακυβεύει τις ίδιες τις βάσεις της ελευθερίας του τύπου και την ελεύθερη άσκηση της δημοσιογραφίας αλλά και της άσκησης του δικαιώματος κάθε πολίτη να το πράττει αυτό. Ε, αυτή η διαδικασία μας ανησυχεί βαθύτατα και θα περάσω στις συστάσεις γιατί περνάει ο χρόνος και να σας πω το εξή. Εγώ θα ήθελα να μιλάμε για ελευθερία της ενημέρωσης και όχι ελευθερία του τύπου. Εσείς είστε κοινοβούλιο και ε, εξορισμού ε, εκπρόσωποι του τύπου και δεν είναι ίδιο ενό επαγγελματικού κλάδου ενημέρωση και πληροφόρηση, ανήκει σε όλου. Για να ανοίξει η συζήτηση. Στη συνέχεια, ε, ακούσαμε να λέγονται πολλά για κανόνες και για οδηγίες. Εμείς δεν διαφωνούμε, αλλά θα προτιμούσαμε να μιλούμε για πρότυπα. Κανόνες, δεν υπάρχει κανονικότητα. Αν μιλάμε για κανονικότητα του τύπου, τότε αρχίζουμε να ανησυχούμε. Επίση, ενθαρρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει κατά κύριο λόγο πολιτικό όργανο. Εσεί δεν είστε δημόσια διοίκηση. Κατανοώ ότι είναι περίπλοκε οι διαδικασίε, αλλά ακριβώ κατά τη δική μας άποψη, είστε η μεγαλύτερη ελπίδα για την ελευθερία του τύπου. Και αυτό θα πρέπει να είναι σε υπερεθνικό επίπεδο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς ε, ε, να ε, εξασφαλίσετε να έχουν την ίδια ελευθερία οι δημοσιογράφοι σε όλες τις χώρες, και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για να επανέλθει σε κάποια βασικά στάνταρ ο κλάδος και το επάγγελμα. Θα ήθελα επίσης να αυξήσετε την επιρροή σας στα εθνικά και τοπικά κοινοβούλια. Ε, ξέρετε όλοι τους βουλευτές της χώρας σας θα πρέπει επιγόντως να εργαστείτε εκεί για να προσπαθήσετε να τους κάνετε να καταλάβουν ότι αυτά που ε, κάνουν ε, είναι πράγματα που δεν επιτρέπονται και υπονομεύουν τα θεσμικά όργανα και τη δική σας αξιοπιστία. Βεβαίως με τα άλλα κράτη-μέλη με τα άλλα θεσμικά όργανα ε, να δείτε τι γίνεται από πλευρά θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη, αλλά αυτό έχει όρια. Κοιτάξτε ε, τα οικονομικά, τις διαφημίσεις. Υπάρχουν και μαφιόζικες ομάδες πλέον που παίρνουν τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιων μέσων ενημέρωσης. Και τέλος θα πρέπει να περάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο φιλόδοξο. Και εδώ συμπεριλαμβάνω και την ίδια μας ευθύνη, την ίδια μας, αν θέλετε, και αδράνεια που αφήσαμε να εξελίσσουν όλα αυτά τα πράγματα, εμείς οι δημοσιογράφοι, και την αδυναμία μας έτσι να ταρακουνηθούμε. Έχουμε το ΕΡΜΑ στην Ευρώπη, το Αριάν, αλλά ε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ε, παραπονιόμαστε για την Google, αλλά δεν έχουμε μηχανή αναζήτησης γνήσια ευρωπαϊκή. Αυτό είναι το θέμα και ε, ίσως το διακύβευμα και ε, δεχομένω και η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο σας να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριο Ολυβία Μπαζίλ. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Βίλεμ Χόσλεϊ που εκπροσωπεί την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Και αμέσως μετά συζήτησης. Συζήτηση και για το δεύτερο και για το τρίτο πάνελ. Ο κύριος Χόσλεϊ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, η ΕΕΔ, ευχαριστεί την Επιτροπή σας για την πρόσκληση. Είχαμε την ευκαιρία το Μάιο φέτος να προβάλλουμε ορισμένες προτάσεις και ε, μαζί με την ε, Επίτροπο κυρία Κρούς και άλλους ευρωβουλευτές γιορτάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ιταλία την 50η επέτειο αυτής της Ένωσης Ευρωπαϊκής Ευρωπαίων δημοσιογράφων και ο καθηγητής κύριος Παπαστάμκος και η επίτοπος κυρία Κρούς δεσμεύτηκαν σοβαρά να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματά μας, διότι βλέπουμε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη, όπως ακριβώς είπε και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ε, είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Θα αναφέρω ε, ε, ε, εν συντομία τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από τη βάση. Η βασική μου προσέγγιση σε αυτά τα προβλήματα είναι. Καταρχάς, συμφωνώ με την κυρία Πέγκη Βάλκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιεί τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Και ο λόγος που δεν το χρησιμοποιεί, ιδίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι επειδή υπάρχει πολιτική ευαισθησία στις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτή η δικαιολογία ούτε καλή είναι ούτε επαρκής. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της και να επιβάλλει ελέγχους δικούς της. Εμείς έχουμε το καλύτερο νομοθετικό σύστημα προστασίας της ελευθερίας έκφρασης και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει πολλές αποφάσεις για την προστασία των πηγών, των δημοσιογραφικών πηγών, για την άρνηση ειδική προστασίας έναντι κατηγοριών συκοφαντικής δυστήμησης για δημόσια πρόσωπα κλπ. κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή νομολογία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σας δίνω ένα, έτσι, μια γεύση των απόψεων της βάσης. Είχαμε γραπτές εξαίσεις από 10 χώρες, συμπεριλαμβάνες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κροατίας, εξαίσεις που έχουν δημοσιευτεί. Και αυτά που λένε σε εκθέσεις, τα παράπονα δηλαδή, τα οποία είναι θα έλεγα σε όλες τις εκθέσεις από τις 20 χώρες που εκπροσωπούνται αναφερόντουσαν στην Ελλάδα και το κίνδυνο βιαίων ε, πράξεων ε, καθημερινού εκφοβισμού και αστυνομικών ε, πράξεων, αστυνομικής βίας κατά δημοσιογράφων στη Ρουμανία και Βουλγαρία ένας πολύ μεγάλος ε, βαθμός ε, δηλητηρίασης των μέσων ενημέρωσης από κατάχρηση εξουσίας από πλευράς ιδιοκτητών η οποία είναι ε, στην αγκαλιά των πολιτικών και της κυβέρνησης και μέσα στα σύνορα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσουν επιτέλους οι νομοθέτες. Στην Κροατία στην Εβδομαδια εφημερίδα Νασιονάλ ε, αναγκάστηκε να κλείσει επειδή υπέστη επιθέσεις πριν από μερικά χρόνια. Οι πράξεις βίας είναι καθημερινές. Ε, στη Βουλγαρία επίσης ακούσαμε να παρεμποδίζονται ε, οι αναφορές στην κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων Όλα αυτά τα θέματα πρέπει επιγόντως να τα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω επίσης να πω και κάτι όσον αφορά το ότι τα παθήματα του παρελθόντος, τα μαθήματα του παρελθόντος δεν χρησιμεύουν ε, στην λύση, ε, τη σημερινή λύση. Δηλαδή το πάσημα δεν γίνεται μάθημα. Ε, έχουμε ενημερωθεί για το εύρος της διαφθοράς σε ορισμένες χώρες και για την οποία δεν έχει γίνει τίποτα. Ανέφερα βεβαίως τις ε, ρήτρες ασφάλειας ε, από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης συγκεντρώσει τεράστια δύναμη όσον αφορά την κατακράτηση ατομικών στοιχείων, ε, Επίση το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ε, δηλαδή αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τη, τη ζωή των πολιτών. Αλλά στο θέμα της διασφάλισης της ελευθερίας ε, φοράει παροπίδες, είναι τυφλή. Παραδείγματο χάρη όταν ο, ο, ο, νόμος για τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ε, ισχυρίστηκαν ότι έχουμε τα μέσα υποπτίας και ελέγχου, ενώ αυτό δεν ισχύει καθόλου. Τα, ε, τον τελευταίο χρόνο η Κομισιόν πάτησε πόδι και μίλησε για την ελευθερία της ε, ενημέρωσης, ελευθερία του τύπου στην Ουγγαρία, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Ε, έγινε μία διάσκεψη 400 δημοσιογράφων και ε, στις Βρυξέλλες οι οποίοι εξέφρασαν τεράστια παράπονα για τη μεταχείριση την οποία υφίστανται. Απαράδεκτη. Ε, επίσης σημειώνω στις, στις σημειώσεις μου θα δείτε διάφορες αναφορές σε διατάξεις και παραγράφους της Συνθήκης Λισαβόνης οι οποίες στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για το αν Ευρωπαϊκή, για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτών των προβλημάτων. Εγώ συμφωνώ όμως με τους άλλους ομιλητές, δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο η νόμη, αλλά είναι η βούληση, η πολιτική που μας πρέπει να μας οδηγεί. Ε, είναι πολύ δύσκολο βεβαίως να βρει κανείς ε, ανεξάρτητους εμπειρογνώμενες να, να αντικρούσουν αυτά τα θέματα. Ε, πρέπει κανείς να κινηθεί ευρύτατα και να ακούσουμε όλες τις φωνές, όπως είχαμε την ευκαιρία σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πλουραλισμού Τύπου και Ελευθερία των ενημέρωσης, του Μέσων Ενημέρωσης έχει παρουσιάσει την πρώτη της έκθεση για τι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα ε, ολόκληρη την παρουσίαση αυτή στο βίντεο και η άποψή μου επί τη βάση αυτής τη παρουσίας είναι ότι και πάλι είναι μια χαμένη ευκαιρία αυτή η έκθεση. Ενδέχεται να είναι μια χαμένη ευκαιρία. Αυτό το κείμενο, από ό,τι ε, βλέπω, δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το δηλητήριο, αυτή τη στρέβλωση που, που γίνεται από την συστηματική κατάχρηση εξουσίας δημοσίων ε, αρχών ε, είναι μία τεράστια στρέβλωση των ελευθεριών, μία έχηση δηλητηρίου από την πλευρά της εξουσίας ε, και το, το θέμα αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Οι συστάσεις της ομάδας υψηλών ε, στελεχών την αναμένουμε και εντυπωσιάστηκα από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Ίδρυμα και την έκθεση του, η οποία λέει, είναι πολύ ενθαρρυντική και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προσφέρει υψηλό βαθμό κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της ελευθερίας του τύπου. Ε, θα παρουσιάσω Έχουμε παρουσιάσει ορισμένε τροπολογίε στο σχέδιο έκθεση. Δεν θα τι παρουσιάσω όλε βεβαίω γιατί τι έχετε γραπτό. Αλλά στο άρθρο 9 πιστεύουμε ότι η Κομισιόν δεν θα πρέπει να αποτελέσει το όργανο για την εποπτεία και την επιβολή ε, κανονισμών ε, και μεθόδων που θα ταιριάζουν σε όλους. Δηλαδή να είναι ένα κουστούμι ραμμένο και κομμένο στα μέτρα όλων. Ε, πρέπει να πιέσουμε και τις κυβερνήσεις και ε, στα κράτη-μέλη και τα θεμελιώδη όργανα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το άρθρο 9 θα πρέπει να λέει ότι καλή ε, την ε, υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων για την καταχείρωση της ελευθερίας στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με το Ίδρυμα Σεμελιωδών Ελευθεριών και των Αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών και έχοντας υπόψη και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, θα μπορέσει να επιβάλλει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει αποτύχει να χρησιμοποιήσει τις ε, ουσιαστικές δυνάμεις που έχει για να διασφαλίσει την συμβατότητα με την συνθήκη της, ε, του, του Συμβουλίου της Ευρώπης παρόλο που θα πρέπει εκ παραλίλου να ε, επιβάλλονται αυτά τα δύο, αυτές οι δύο σαμελιώδεις κανονισμοί για την προστασία των δημοσιογράφων. Ε, νωρίτερα φέτος η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου ε, της Ευρώπης ε, έκανε μια αρκετά σαφή δήλωση ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, διορατικότητα κλπ. και Ε, και ότι θα δημιουργήσετε εργαλεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρειάζεται. Ε, αυτά δεν είναι επαρκή. Διεθνώ, η ελευθερία του, των μέσων ενημέρωσης όχι μόνο δέχεται επιθέσεις αλλά καταστρέφεται σε πολλές χώρες. Πριν από 10 μέρες στο Λονδίνο ε, είχα διοργανώσει μία συνάντηση 60 ηγετικών συντακτών και δημοσιογράφων σε ένα κτίριο του BBC. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εκδώσαμε μία δήλωση του Λονδίνου η οποία θα υποβληθεί ε, στις 22 Νοεμβρίου στην συνάντηση που θα γίνει στα πλαίσια του ΟΗΕ και ο Διευθυντής Διεθνών Ειδήσεων του BBC είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα προσκόμματα, οι φυσικές ε, απειλές, ε, σωματικές πράξεις βίας και εμποδίζουν, είναι τεράστια εμπόδια αυτά για την ελεύθερη αναφορά ε, των ειδήσεων και αυτού που, αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι σε καλύτερη θέση από ότι άλλα μέρη του κόσμου, ε, όπως έχει δημοσιευθεί στην έκθεση του ΟΗΕ. Ε, στο σημείο 19 που λέει ότι η Ευρώπη είναι μία από τις χειρότερες οντότητες παγκοσμίως για την προστασία το, του τύπου. Και πραγματικά πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Ο Πρόεδρος, ε, παρακαλώ να συνεργαστούμε διότι έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Οι ομιλητές ε, των πάνελ ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους ε, και δεν έχουμε καιρό, λέει η κυρία Βέμπερ. Ε, στον πρόεδρο. Ε, Τέλο πάντων, ένα λεπτό, ενάμιση σε όσους θέλουν να παρέμβουν και μετά να απαντήσουν οι πανελίστες. Παρακαλώ να είστε τηλεγραφικοί. Η κυρία Μόρβαϊ. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι και οι διεθνείς δημοσιογράφοι με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν θεσμικό όργανο. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ελευθερία του τύπου και την υποχρέωση και το δικαίωμα μάλλον που έχουν οι πολίτες για ενημέρωση. Γιατί το ρωτάω γι' αυτό. Διότι η κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι είναι θυμωμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί λένε ότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχει ένα ανήθικο λόμπι, θέλουν περισσότερες, ε, ε, περισσότερη διαφάνεια, θέλουν ακριβώς όπως και στα κράτη-μέλη να υπάρχει διαφάνεια για την ε, λήψη των πολιτικών αποφάσεων, να είναι υπόλογοι οι πολιτικοί, να παρακολουθούμε δηλαδή τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των πολιτικών οργάνων. Ακούμε συχνά ε, κριτική για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Αλλά ας πούμε για την Ουγγαρία το ακούμε συνέχεια. Αλλά δεν ακούμε ε, καμία κριτική ε, για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαινόμενα αυτά γιατί δεν ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Ο κύριος Μπορσελίνο, 1,5 λεπτό. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία περίπτωση πολύ ιδιαίτερη στην Σικελία, στην Ιταλία. Η Σικελία είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση σε μία χώρα που δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Οχτώ δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι απειλούνται ακόμα και σήμερα και προστατεύονται αυτή τη στιγμή η ασφάλεια των δημοσιογράφων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι θέμα αστυνομίας και μόνο. Η Ένωση Δημοσιογράφων, η Ομοσπονδία Δημοσιογράφων πώς αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ο κύριος Ρούτσας. 1,5 ε, όχι δύο λεπτά για να πάρω και το μισό λεπτό της κυρίας Μπορσαλίνο. Μία δήλωση, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αλλά θα ήθελα να πω όμως ε, ε, λίγα λόγια για την κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις. Ε, ε, κατά την άποψή μου η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κοινωνική, είναι και κρίση αξιών και κρίση δημοκρατίας και ο ρόλος των ρόλων εδώ είναι ζωτική σημασία για την κατάσταση. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές. Ε, το σύστημα των ΜΜΕ στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια πάρα πολύ στενή σχέση ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτικό κόσμο και τα ΜΜΕ ε, αυτά τις τελευταίες εβδομάδες ε, είμαστε μάρτυρες ε, πολύ ανησυχητικών εξελίξεων όταν η κυβέρνηση παρεμβαίνει χωρίς απροκάλυπτα στην, στα ΜΜΕ. Ακούσατε την σύλληψη του δημοσιογράφου του κ. Βαξεβάνη, διότι δημοσίευσε την περίφημη λίστα. Υπάρχουν πολιτικές ε, κόβονται μάλλον κόβονται εκπομπές ενημέρωσης στην ε, ελληνική τηλεόραση διότι δεν παρουσιάζονται τα πράγματα του δημοσιογράφους έτσι όπως τα θέλανε οι κοινοί κυβερνήσεις. Ε, μία τελευταία παρατήρηση, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, ο, ο σκοπός μου δεν είναι να κατηγορήσω τη χώρα μου και ιδίως τώρα που περνάμε αυτή την κρίση, όμως πιστεύω ότι η κρίση αυτή στην Ελλάδα είναι και μια ευκαιρία να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή, να δημιουργηθεί μια νέα Ελλάδα και ο ρόλος των μέσων είναι ζωτικό. Εάν δεν θέλουμε οι θυσίες των ε, Ελλήνων πολιτών να είναι μάτες, ε, θα πρέπει να γίνει κάτι ουσιαστικό, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρξει μια νέα Ελλάδα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και όχι ερωτήσεις. Ε, αλλά τέλος πάντων, και ούτως ή άλλως και ερωτήσεις, ποιος θα τις απαντήσει, αυτό δεν έχουμε χρόνο. Ε, ήθελα να πω ότι ακούστηκαν πολλά σχόλια ε, γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται όχι μόνο σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε ε, να, από τα γραφειοκρατικά προβλήματα ή διλήμματα αλλά ένα άλλο σημαντικό για μένα μήνυμα ήταν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πολιτικό σώμα και άρα θα πρέπει να λειτουργούμε και να δρούμε σαν πολιτικό σώμα που θα πρέπει να ενθαρρύνει να προχωρούμε μπροστά. Η κρίση δεν είναι μια δικαιολογία. Η κρίση δημιουργεί νέες δυσκολίες και νέες προκλήσεις για όλους μας και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο την κρίση και να εστιάσουμε στην κρίση. Ε, ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός επίσης και η, η εντολή μας πρέπει να διευρυνθεί και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μην χάσουμε την ευκαιρία με την έκθεση αυτή, να μην χάσουμε κι άλλη μια ευκαιρία. Αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Το ένα είναι ότι πολλές, πολλοί από τους ομιλητές ασφε, αναφερθήκανε στον ρόλο του κράτους και στην κρατική διαφήμιση. Και ο κύριος Δράγκομιρ και ο κύριος Χόρσλι ε, μίλησε επίσης και για τους δημόσιους αξιωματούχους που χρησιμοποιούν ε, κρατικούς πόρους ε, ο Πρωθυπουργό μας, παραδείγματο χάρη, δεν ήθελε να μιλήσει ε, στην, σε μια ερευνητική επιτροπή του Κοινοβουλίου ε, γιατί έπρεπε να μιλήσει για τη χρηματοδότηση μιας εφημερίδας κτλ. Εγώ ρωτώ Ούτω ή άλλω στην Αυστρία αλλάξαμε την νομοθεσία και καταστήσαμε σαφέ ότι κανένα υπουργό, κανένα δημόσιο ε, ε, λειτουργό δεν μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιε φωτογραφίε, τέτοιου είδου ε, διαφημιστικέ φωτογραφίε. Και αυτό είναι μία πρόοδο. Επίση. Εξεπλάγει πάρα πολύ. Ήμουν το πρωί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών και ψηφίσαμε εκεί και ήρθε ένα mail από το δικό σας γραφείο χτες και μας ζητούσε να απορρίψουμε κάποιες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με στερεότυπα με βάση το φύλλο. Και Δηλαδή ότι να θεωρούνται οι γυναίκες αντικείμενα, να προβάλλονται έτσι και να ε, ε, ζητήσουμε να επιταχυνθεί ε, θέλαμε η κείμενη νομοθεσία κατά των στερεοτύπων και ήρθε το γραφείο σας και μας ζητούσε να τα απορρίψουμε. Ε, αυτό είναι μια ηθική πίεση που δεν μας αρέσει εμάς ε, τους βουλευτές και χρειάζονται και τα μέσα εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση. Γιατί μας ζητάτε να μην ψηφίσουμε τέτοιες σημαντικές τροπολογίες, η κυρία Σαρζεντίνη. Ε, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω ε, πραγματικά με μεγάλη ευκολία ε, από εκεί που σταμάτησε η κυρία Τσέκ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ρούσα. Άκουσα αυτή την έκκληση των εκδοτών εφημερίδων να μην υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Εδώ και χρόνια τα ακούω αυτά για την πολυφωνία στα μέσα. Και Πώς απαντάς αυτά που βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις εταιρείε στον πληθυντικό του Ρούπερτ Μέρντοκ που καταχρώνται σαφώς της ε, οικονομικής τους ισχύω. Και δεν είναι κατά ανάγκη ισορροπημένη η ενημέρωση και τα μέσα, τα μίντια του ομίλου Μέρντοκ. Και κάνετε και άλλη πρόταση τώρα Ε, μια πραγματική πρόταση, όχι αυτορύθμισης, ουσιαστική ε, για προστασία της ελευθερίας και της πολυφωνίας στον τύπο. Ευχαριστώ κύριος Προτασίεβιτς. 1,5 λεπτό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, πρόεδρε. Εξ όσων κατάλαβα, ακούσαμε και τον κύριο Μπαζίλ και τον κύριο Χόσλι να μας λέγουν ότι ε, το θέμα της συγκοφαντικής δυσφήμισης ε, κατά των υψηλών αξιωματούχων και των ε, αρχηγών κρατών είναι βασική πρόκληση. Και τι ρόλο καλείται εκεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ρόλος με ρύθμιση, με πρόταση για αλλαγές και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα τελικά. Ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ακούσαμε ε, τον καημό των καημένων των δημοσιογράφων και των διοκόμενων εφημερίδων, ότι θα πρέπει να μην έχουν περιορισμούς και συμφωνούμε ότι χρειάζονται προστασία από καταστολή της κυβέρνησης ή ε, της νομοθετικής εξουσίας. Αλλά πώς προστατεύονται τα προστάτευτα θύματα του τύπου. Ακούσαμε ε, πώς χρηματοδοτούνται ε, και ότι δεν μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν συγκεκριμένους τίτλους, συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα και ε, το θέμα της οικοφαντική δυσφήμισης μπορεί να το αντιμετωπίσουν μόνο οι πλούσιοι. Τα κρατικά μέσα ε, που είναι εχέγγυα αμεροληψίας μπορούν να αντιμετωπίσουν τους βαρώνους του ιδιωτικού τύπου, αλλά στο BBC έχουμε κατάλογο ευνοουμένων που έχουν ε, απεριόριστη πρόσβαση και κάποιων άλλων δαιμόνων που τους ε, αποκλείεται κάθε πρόσβαση και ε, κάνουν τους κανόνες τους και τους ακολουθούν. Και τελικά αυτό που εξισώνει τους πάντες είναι το διαδίκτυο. Ε, νωρίτερα φέτος η Ευρωπαϊκή ε, Επίτροπος Ρέντινγκ πρότεινε να διωχθεί νομικά η ιστοσελίδα του Ολλανδικού Κόμματος Ελευθερίας γιατί δεν της άρεσε το περιεχόμενό της. Ο Πρόεδρος, πιστεύω ότι τέθηκε μία ε, σαφής ερώτηση προς τον κύριο Ράσταλ, όμως όλοι έχουν τη δυνατότητα να, να απαντήσουν, ε, δεδομένου ότι είχαν συμμετέσχον στο δεύτερο και τρίτο πάνελ. Άρα λοιπόν δίνω το λόγο καταρχάς στην καθηγήτρια κυρία Φάλκε. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ωραία. Ο κύριος Ντράγκομιρ. Ευχαριστώ. Απλώς θέλω να απαντήσω όσον αφορά τα δίκαια κριτήρια για την κατανομή των κρατικών διαφημίσεων της κρατικής προβολής. Αυτό πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με πιο περίπλοκα θέματα ε, όσο παραδείγματος χάρη της συστάσεις ε, για την ε, ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. Τώρα όσον αφορά την κατανομή των κρατικών, της κρατικής προβολής ή διαφήμισης, το πρώτο μέτρο θα ήταν να επιβληθεί διαφάνεια, διαφάνεια και δημοσίευση των πιστώσεων που χρησιμοποιούνται πρόσβαση και πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Δεύτερο βήμα είναι η υιοθέτηση που δεν έχει συμβεί σε πολλές χώρες. Μηχανισμοί, δηλαδή δίκαιες κατανομής της κρατικής διαφήμισης πρέπει να βασίζονται σε ξεκάθαρα κριτήρια κατανομής και σωστής διαχείρισης και τρίτον τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, οι εθνικές ελεγκτικές αρχές, τα ελεγκτικά ναι, συνέδρια, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να επιβάλλουν δίωξη ή νομικά μέτρα ή κυρώσεις αν θέλετε όταν δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάλτερ, έχετε κάτι να προσθέσετε με τα αυτά που είπε ο κύριος Ντράγκομι. Όχι, ευχαριστώ, με κάλεψε. Ο, η κυρία Φρανκ. Όχι. Ο κύριος Ράστα. Ευχαριστώ. Μια που έχω δύο ερωτήσεις, ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω με μία πρόταση για κάθε ερώτηση. Καταρχάς, κυρία Λούνιτσεκ, για τη δική μας παρέμβαση και τη συζήτηση της δοτερότητας ε, των φύλων. Είναι σαφές ε, ότι εμείς ε, δεν θέλουμε καμία πολιτική ρύθμιση του τύπου. Δεύτερον, η ατυχής κατάσταση στις, στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας από τους συναδέλφους μας ε, παρεύει τον νόμο. Αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Ε, βεβαίως, αλλά η αυτορύθμιση στο Ενωμένο Βασίλειο είναι υπερβολικά δύναμη, όπως αποδεικνύει αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε με αυτόν τον δημοσιογράφο. Και τέλος, σας προτείνω να ξαναδιαβάσετε, να ξανακούσετε την ομιλία του κυρίου Χόρσλι, ο οποίος μας είπε ότι η Ευρώπη έχει το πιο ισχυρό δίκτυο πρόστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο αυτό να κοιτάξει να επιβάλλει τους σωστούς κανόνες και όχι μόνο και αποκλειστικά μέσω των νόμων. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και το τρίτο πάνελ, ο κύριος Κιόνικ, ευχαριστώ. Όσον αφορά την Ουγγαρία και το επιχείρημα ότι δεν επικρίναμε άλλες χώρες, δεν συμφωνώ. Οι ρηπόρτες χωρίς σύνορα έχουν κατακρίνει και άλλες χώρες δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, έχει έχει υπάρξει επιστοχώρηση προστασίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση όταν επισκεφθήκαμε την Ουγγαρία πέρσι αλλά και η Ρουμανία και η Μακεδονία που μπορεί να περαστούν από αυτή την Ουγγρική νομοθεσία όλοι οι νομικοί εμπειρογνώμονες για την ελευθεριοτυπία μου λένε ότι το ουγγρικό παράδειγμα αρχίζει και διαρρέει πλέον και έχει επιπτώσεις και σε γειτονικέ χώρες δεν βλέπω πώς η Ευρώπη μπορεί με καλό τρόπο να χειριστεί το θέμα της Τουρκίας, δεδομένου, αν δεν έχει την ηθική βάση, το, την ηθική πλατφόρμα από την οποία μπορεί, μπορεί να ομιλεί και πιστεύω ότι θα ακολουθηθεί ένας παρόμοιος δρόμος όπως της Ουγγαρίας, ο κύριος Μπαζίλ. Ναι, πάρα πολύ σύντομα έγινε μια ερώτηση αν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση. Απάντηση όχι, σαφέστατα. Σα το είπα. Οπισθοδρομούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ω μη κυβερνητική οργάνωση και κάτοχοι του βραβείου Ζαχάροφ θα καταπολεμήσουμε όλα αυτά που τώρα προπτύνονται στην Ένωση. Ε, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι γίνεται πίσω από τις πόρτες της Ευρώπης και γιατί. Ε, διότι δεν εργαζόμαστε. Ε, Έχουμε πολύ σοβαρούς δημοσιογράφους, ε, αλλά και, και δημοσιογράφους που κάνουν λιγότερο καλά τη δουλειά τους, όπως όλοι οι κλάδοι. Αλλά παράγεται πολύ μεγάλο νομοθετικό έργο και είναι πολλά τα θέματα στην Ευρώπη και το θέμα δεν είναι ότι έχουμε κρυφή ατζέντα, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα καλύψουμε όλα. Στην Ιταλία η κατάσταση των δημοσιογράφων είναι πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι στην Ιταλία έχουν προστασία. Για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα τη ελευθεροτυπία στην Ελλάδα ήταν ότι βασίστηκε σε μια χρηματοδότηση τελείω ε, χωρίς καμία αξιοπιστία η χώρα και κατέρευσε αυτό μετά από οικονομική κρίση. Αυτό είναι παράδειγμα, διδάσκεται στις σχολές στο μέλλον. Και για τη Βουλγαρία το θέμα είναι η διαχείριση ε, των ε, εταιριών διαφήμισης, γιατί ε, και να, γίνεται ένας κατάλογος να καταγράφονται που πηγαίνουν τα χρήματα, όπως κάνει ο ιδιωτικός τομέας και στο δημόσιο και όχι να αρνείται ο, ο υπουργός να έρθει να καταθέσει. Δεν μπορώ σε 60 λεπτά τώρα, τελευταίος ομιλητής, το θέμα για την Ιταλία που τέθη και τους δημοσιογράφους που ζουν στο φόβο ή που δολοφονούνται. Αυτό υπογραμμίζει απλούστατα το γεγονός ότι η δυνατότητα των δημοσιογράφων να ενημερώνουν ε, το κοινό είναι θέμα θεμελιώδους ε, ε, κράτους δικαίου και αν εκφοβίζονται οι δημοσιογράφοι και αναγκάζονται να αυτολογοκρίνονται ή να κρύβονται, κοιτάξτε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό σε μια χώρα και θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρώπη γενικότερα. Το μεγάλο ζήτημα εδώ ε, της έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμπεριφορά του τύπου έχει απόλυτο δίκιο ε, ο, ο, ήταν πραγματικά αποτρόπε αυτή η συμπεριφορά ε, και πονίδιστη ε, και ικτροί και χιλιάδες άνθρωποι ε, μπορούν να δουν τη ζωή τους να καταστρέφεται από ένα ιδιοκτήτη εφημερίδα σκανδαλοθυρική. Αυτό συγκλώνησε το σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω ότι κατάλαβαν και οι δημοσιογράφοι και οι εκδότε ότι δεν μπορούν να είναι καρτέλ θα πρέπει να είναι υπόλογοι στο κοινό με τρόπο πιο πιστικό. Δηλαδή η νέα δομή, ο νέος θεσμός που θα ακολουθήσει τον παρόντα θα προσπαθήσει να το κάνει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δημοσιογράφοι, όχι η αστυνομία, αποκάλυψαν ε, το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χρειάζεται ελεύθερος τύπος για να το κάνει η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κοινού και ούτε η πολιτική όταν μία από τις ε, εταιρείες των ε, media έγινε πανίσχυρη αυτό το θέμα της συκοφαντικής δυσφήμισης, ε, αυτό το θέμα και ο βαθμός του προβλήματος, πώς χρησιμοποιείται αυτός ο νόμος περί συκοφαντικής δυσφήμισης. Ακούσαμε την Τούνια Μιγιάτοβιτς προηγουμένως ότι ποινικοποιείται ε, και υπάρχει ακόμα ε, ποινικό αδίκημα αυτό το θέμα και είναι καθημερινό ψωμοτήρι πολλών δημοσιογράφων της Ένωσής μου. Εμείς Χαιρόμαστε για τη στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα της Επιτρόπου κυρίας Κρούς, η οποία είπε ξεκάθαρα ότι φοβάται και είναι απρόθυμη να προχωρήσει σε κάτι που μπορεί να αποδειχτεί μπούμεραγκ για την ελευθερία του τύπου. Ε, αυτό είναι σωστή προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα όλοι οι δημόσιοι θεσμοί και οι πολιτικοί θα πρέπει να σταματήσουν να προστατεύουν ε, τους δικούς τους πολιτικούς και τη δική τους πολιτική δράση. Θα πρέπει να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι τα θεσμικά όργανα εργάζονται υπέρ της γνήσιας ελευθερίας του τύπου. Και τέλος, ε, ε, τα δημόσια ε, όργανα και θεσμοί όπως η EBU και οι άλλοι θεσμοί έχουν ρόλο εδώ να παίξουν και θα πρέπει να δώσουν ήδη το παράδειγμα διαφάνειας στο σπίτι μας στην Ευρώπη, όχι μόνο έξω και ο διαγωνισμός της Eurovision φέτος στο Αζερβαϊτζάν δεν έκανε καλό στα δημόσια θεσμικά μας όργανα και τους θεσμούς μας. Χρειαζόμαστε και επαγρύπνηση και διαφάνεια και από πλευράς πολιτικών, όχι μόνο το μέσων ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος, όλους τους ομιλητές μας και τα μέλη του πάνελ. Ξέρουμε ότι έχουμε καθυστερήσει πολύ. Ζητούμε συγγνώμη ε, που σας πιέσαμε στο τέλος. Έτσι συμβαίνει συνήθως στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για τις προσπάθειες που κάναν να ε, μειώσουν τις ε, ρουσιάσεις και έμειναν μέχρι τέλους για να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Και τώρα Πρέπει να ανακοινώσω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. 20 Νοεμβρίου αντί της 8ης, 20 Νοεμβρίου λίγη προθεσμία το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ και πάλι και τώρα ακολουθούν οι συντονιστές.